Meine Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας καλωσορίσω εγκαρδιότατα. Παρακαλώ να κάτσετε στις θέσεις σας. Το πρώτο πάνελ δεν είναι καν πλήρες εδώ. Και ο ίδιος το έζησα. Οι αφήξεις στο αεροδρόμιο είχαν καθυστέρηση μέχρι και μία ώρα καθυστέρηση. Αλλά θα αρχίσουμε παρόλα αυτά. Το θέμα του εργαστηρίου σήμερα είναι η επιπτώσεις της κρίσης της ΜΜΕ. Ένα θέμα ιδιαίτερα σημαντικά για την Ευρώπη και για την εργασία μας. Γιατί ξέρουμε όλοι ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ε, σπονδυλική στήλη της ε, ευρωπαϊκής οικονομίας. Εκείνοι δημιουργούν θέσεις απασχόλησης. Εκείνοι είναι πιο καινοτόμοι και δημιουργικοί και συμβάλλουν έτσι στο οικονομικό αποτέλεσμα της Ευρώπης. Αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως αποδεικνύουν και ε, δημοσκοπήσεις, είναι εκείνες που πλήττουν ιδιαίτερα από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Έχω εδώ μία αξιολόγηση Euroshambo που έκανε μία δημοσκόπηση ανάμεσα στα μέλη του και από την οποία προέρχεται ξεκάθαρα ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, διαμαρτύρονται γιατί έχει επιδεινωθεί, έχουν επιδεινωθεί οι όροι για την δανειοληψία και ότι έχει επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο οι τρόπος με τον οποίο πληρώνουν ε, από το δημόσιο και γι' αυτό υπάρχουν απώλειες και αυτές οι επιχειρήσεις κατά 30% το 1 τρίτο δηλαδή είπανε ότι θα μειώσουν προσεχώς τις επενδύσεις τους. Δεν μπορούν να τηρήσουν το σημερινό επίπεδο. Το 60% των επιχειρήσεων αυτών, μόνο το 60% λέει ότι θα παραμείνει η απασχόληση στο επίπεδο που έχουν. Και το 20% κάθε πέμπτη επιχείρηση δηλαδή θεωρεί ότι θα μειωθεί το επίπεδο απασχόλησης. Είναι πάρα πολύ κρίσιμη λοιπόν η κατάσταση και αυτό χαίρομαι που έχουμε μεταξύ μα εμπειρογνώμονε που θέλουν να συζητήσουν αυτό το θέμα. Έχουμε κατανείμει την, το εργαστήριο αυτό σε δύο τμήματα. Καταρχήν θέλουμε να συζητήσουμε πώ. Ποιο ήταν ο αντίκτυπο τη κρίση μέχρι στιγμή στι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Έχω τρει εμπειρογνώμονε. Έχετε τα βιογραφικά του ε, σημειώματα, δεν θα ήθελα να αναπτύξω. Έχουμε τον Αντώνιο Σαράιβα από την Πορτογαλία πρόεδρος του Εθνικού Σώματος Εκπροσώπησης της ε, Προγαλλικής Βιομηχανίας, την Μαρία Νόβουεκ, που εργάζεται στο European Microfinance Works στο Παρίσι. Και έχουμε τον Πόντους Μπράουνχερμ, ο οποίος έρχεται τώρα, που είναι από την Σουηδία. Και στο δεύτερο τμήμα θέλουμε να συζητήσουμε προτάσεις ποιες είναι οι πολιτικές αποφάσεις που θα μπορούσαν ίσως να ληφθούν υπόψη για να αντιμετωπιστούν αυτές οι δυσκολίες. Του συμμετέχοντες στο δεύτερο πάνελ θα σας παρουσιάσω μετά. Όπως συνήθως θα δώσουμε στους τρεις εμπειρογνώμονες καταρχήν το λόγο, παρακαλώντας τους να μιλήσουν ο καθένας 10 λεπτά περίπου και κατόπιν θα έχουμε τη δυνατότητα να υποβάλουμε ερωτήσεις. Πριν περάσουμε στο δεύτερο πάνελ, θα ήθελα καταρχήν να σας δώσω το λόγο. Καλώς ορίσατε και σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε εδώ μαζί μας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Θεωρώ πως αυτό το σεμινάριο έχει θεμελιώδη σημασία για τη μελλοντική ζωή του επιχειρηματικού κόσμου. Καταρχήν, η κρίση επηρέασε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτό θα δούμε πώς έγινε. Και δεύτερον, πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, δηλαδή που κατευθυνόμαστε για το μέλλον. Μου ζητήθηκε να προσεγγίσω το πρώτο θέμα, να κάνουμε δηλαδή μια διάγνωση για την επιχειρηματική κατάσταση αυτή τη στιγμή, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να αναλύσουμε τα βασικά προβλήματα που αυτές αντιμετωπίζουν στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα από αυτά τα προβλήματα επιδεινώθηκαν ιδιαίτερα μέσω της οικονομικής, χρηματοπιστωτικής και κοινωνικής κρίσης, την οποία αντιμετωπίζει ολόκληρος ο κόσμος. Αρχικά θα μιλήσω για τον επιχειρηματικό ιστό της Πορτογαλίας, μετά για τον αντίκτυπο της κρίσης και τέλος θα αναφερθώ σε κάποιες από τις δυσκολίες που ιδιαίτερα αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, στην επιδείξη των στόχων τους. Η πορτογαλική επιχειρηματική δομή ε, η καινοτομία και την που εισήχθη το 2007 οδήγησε στην Πορτογαλία το 2008 να υπάρχουν 372.000 ε, εταιρείε, δηλαδή 370 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και απασχολούσαν 2.800.000 ε, ε, ε, υπαλλήλους. Πρόκειται για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κυρίως για πολύ μικρές επιχειρήσεις. Κάθε φορά όλο και περισσότερες είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτές είναι υπεύθυνε ε, για δύο από τις τρεις επιχειρήσεις που υπάρχουν. Στην Πορτογαλία, σύμφωνα με τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, παρατηρούμε ότι υπάρχουν περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανακάτοικο σε σχέση με τις 27 υπόλοιπες χώρες της Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε μόνο και αποκλειστικά με τις μικρομεσαίες αγνοώντας τις μεγάλες επιχειρήσεις. Εμείς θέλουμε και ελπίζουμε ολόκληρη η οικονομία να ανακάμψει και οι μικρομεσαίες μαζί της. Είναι ωστόσο ε, πολύ σημαντικό να δούμε τις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και φωτίζοντας τα, τα, τα εμπόδια Δημιουργώντα καλύτερε προποθέσει για τη δημιουργία του, την ανάπτυξή του και την πρόοδό του. Ποιο είναι ο αντίκτυπος της κρίσης. Με την ε, χρηματοπιστωτική κρίση που ξέσπασε το 2008 υπήρξε μια μεγάλη, ένας μεγάλος αντίκτυπος σε όλα τα επίπεδα, το οικονομικό και της απασχόλησης. Στην Πορτογαλία η ανάπτυξη της οικονομίας το 2008 καθορίστηκε από την εξωτερική κατάσταση που ήταν ιδιαίτερα δυσμενής και ξεκίνησε αυτό από το 2007. Ο αντίκτυπος οικονομικής κρίσης που επιδίνωσε ε, αρνητικές τάσεις που ήδη υπήρχαν. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Εξωτερικού Εμπορίου της Πορτογαλίας, το 2009 υπήρξαν τέτοιες ε, επιπτώσεις που οδήγησαν στην μείωση του PIB με μεταβλητή μηδενική για τον όγκο του έναντι του 1,9 το 2007. Ε, το 2007. Υπήρχε επίσης σε μείωση των αγαθών και των υπηρεσιών κατά 0,5% και η μείωση των επενδύσεων ήταν πολύ σημαντική και το 2008, μείον 1,1% ενώ είχε αυξηθεί κατά 3,7% το προηγούμενο έτος. Το βασικό εθνικό μας Ινστιτούτο της Στατιστικής διαπίστωσε ότι το 2008 το 2009 και το 2010 μας έδωσαν τα στοιχεία που μπορείτε να δείτε στον πίνακα, ε, στην ε, διαφάνεια που έχουμε. Δεν βλέπουμε πότε, έγινε, ε, πότε ήταν η αρχή της κρίσης μέσω των στοιχείων. Μια μεγάλη οικονομική κρίση ωστόσο ήδη μενόταν σε εθνικό επίπεδο στην Πορτογαλία με πολύ σοβαρές οικονομικές συνέπειες που εκφράζονται στο, με τον αριθμό των επιχειρήσεων που πτώχευσαν καθώς και με τον αριθμό των ανθρώπων που απολύθηκαν. Πολύ μεγάλη αύξηση της ε, ανεργίας, καθώς και μείωση των εσόδων των οικογενειών και άρα και συρρήκνωση της κατανάλωσης. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις ε, είναι, γενικά, είναι γενικές και γίνονται αισθητέ περισσότερο στα πιο αδύναμα στοιχεία της κοινωνίας αλλά και των επιχειρήσεων. Όσον αφορά τις μικρομεσαίες, το πιο ευάλωτό τους μάλλον σημείο ε, είναι οι, μικροί τους, οι μικρές τους διαστάσεις και οι λιγοστές δυνατότητες ανταγωνιστικότητας. Έχουν δυσκολίες να χρηματοδοτηθούν, έχουν μεγάλες δυσκολίες όσον αφορά τα διοικητικά τους καθήκοντα, έχουν μεγάλε δυσκολίε όσον αφορά την αγορά εργασία ή χρηματοδότηση. Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητε όσον αφορά την γενικευμένη μείωση των ε, πλαφών. Όπω ε, είναι γνωστό, η πρόσβαση στι πιστώσει έγινε ακόμα πιο δύσκολη και το κόστο ήταν ακόμα πιο ε, αυξημένο. Οι μικρομεσαίε επιχειρήσει αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλε δυσκολίε λοιπόν για πιστώσει σε όλε τι φάσει τη ζωή του και όχι μόνο στην αρχή καμία δεν είχε επαρκή έσοδα ώστε να μπορέσει να πάρει ένα παραδοσιακό τραπεζικό δάνειο. Οι μικρομεσαίες λοιπόν έχουν να αντιμετωπίσουν και άλλα εμπόδια γιατί έχουν πρόβλημα να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Το ίδιο όταν έχουν να αντιμετωπίσουν μια διαδικασία μετατροπής ή μεταρρύθμισης ε, και έχουν, ε, προσκρούν πάντοτε σε δυσκολίες χρηματοδότησης. Τώρα, πέρα από την πρόσβαση στις πιστώσεις υπάρχει ένα επιπλέον βάρος, ένα επιπλέον φόρτος, είναι το κόστος δηλαδή το οποίο πρέπει να φέρουν γιατί οι εγγυήσει που απαιτούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από αυτές τις επιχειρήσεις συνήθως είναι τόσο, τόσο μεγάλες που είναι αδύνατον να τι φέρει μια μικρομεσαία επιχείρηση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν να μην υπάρχει πραγματικός αντίκτυπος και να φτάσουν πραγματικά χρήματα και η αρρωγή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αυτό λόγω των, όλων αυτών των αιτίων που σας εξέθασα. Τώρα, αυτό που είναι πολύ σημαντικό για τα βραχυπρόθεσμες, τις βραχυπρόθεσμες πιστώσεις, που είναι πολύ σημαντικές για τις εμπορικές συναλλαγές, οδηγεί στο να μην μπορούν να δανειστούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να χάνουν τους, ε, πολι... Ε, τους πελάτες τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται σε μια κατάσταση ακόμα πιο ευάλωτη οικονομικά. Για παράδειγμα στην Πορτογαλία στο δεύτερο τρίμηνο του 2008 η μέση προθεσμία πληρωμής της κεντρικής ε, ε, δημόσιας διοίκησης ήταν περίπου ε, 300 ημέρες με ε, maximum 1900 ημέρες. Ε, τότε γινόταν η καταβολή των ε, ποσών. Κανονικά έπρεπε αυτά όλα να γίνονται εντός 100 ημερών. Αυτό σημαίνει το, ε, ότι ακόμα και τα νοσοκομεία είχαν δυσκολίες στο να καλύψουν και να πληρωθούν. Είναι τόσο μακρές οι προθεσμίες, οι οποίες πραγματικά θέτουν υπό αμφισβήτηση την επιβίωση όποιον θέλει να παραμείνει ανεξάρτητος επαγγελματίας. Επίσης οι επιχειρήσεις πολύ συχνά έπρεπε να πληρώσουν το ΦΠΑ για συναλλαγές που έχουν κάνει μέσα στο ίδιο τους το κράτος πριν να έχουν ε, λάβει οποιαδήποτε ανταμοιβή για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Τώρα, ποια είναι η διοικητική πλαισίωση στην Πορτογαλία. Αυτό αποτελεί ένα από του τομεί που είναι οι πιο δύσκολοι και καθορίζουν τι μικρομεσαίες επιχειρήσει και την ανταγωνιστικότητά του. Θα τονίσω κάποιε πτυχέ για τη δημιουργία και τη μετατροπή και για τη σύσταση μιας επιχείρησης είναι πολύ γραφειοκρατική, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που τόσο όσον αφορά την οικονομική επιβάρυνση, όσον αφορά και τη διοικητική. Είναι ιδιαίτερα περίπλοκη η διαδικασία για τη δημιουργία μια νέα ε, επιχείρηση. Υπάρχουν δυσκολίε κατανόηση, ε, διοργάνωση, πέρα από το κόστο που σημαίνει η απόκτηση νέου software που θα επιτρέπει να αντιμετωπίσει κανεί ε, αιτήματα που είναι νομοθετικά επιβαλλόμενα. Η λειτουργία των δικαστηρίων δεν δυσχεραίνει την ε, διαδικασία κάλυψης των πιστώσεων. Ε, Judicial de conflitos não se encontra suficientemente generalizados e desenvolvidos para constituir uma solução. Γενικά έχουν αναπτυχθεί, ε, πρέπει να αναπτυχθούν συστήματα που να διευκολύνουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι πολύ περίπλοκη κατάσταση δεν υπάρχει επαρκή ενημέρωση και δεν υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα. Στι αγορέ υπάρχουν ακόμα πολλά εμπόδια ανάμεσα στα κράτη-μέλη, πράγμα το οποίο δυσχεραίνει την ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Δεν υπάρχει επαρκής γνώση, αμοιβαία γνώση, πράγμα το οποίο επιδεινώνει την παροχή των υπηρεσιών. Η δημιουργία ενώ μια μικρομεσαία επιχείρηση σε μια χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να γίνεται με μια εύκολη επιχειρησιακή διαδικασία. όπως ας πούμε για την Ευρωπαϊκή Ιδιωτική Επιχείρηση. Θα ολοκληρώσω κύριε Πρόεδρε. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, όπως είπαμε, ε, τιμωρούνται από τις διαδικασίες που ισχύουν αυτή τη στιγμή. Οι προδιαγραφές που ισχύουν δεν λαμβάνουν υπόψη αρκούντως τις δυσκολίες αυτών των επιχειρήσεων. Υπάρχουν πάντοτε παραδείγματα ε, πολλές δυσκολίες σε σχέση με την νομική πλαισίωση, την διοικητική και την χρηματοπιστωτική πλαισίωση. Και τα εμπόδια που τίθενται από διάφορες χώρες και που αποκαλύπτονται με διάφορους τρόπους, δασμολογικούς και μη δασμολογικούς, περιορισμούς ποσοτικούς, πρακτικές dumping, εμπορικές, κοινωνικές, ακόμα και περιβαλλοντικό dumping. Θυμίζω πως αυτή η κατάσταση επιδεινώνεται και από το γεγονός ότι αυτές οι επιχειρήσεις μάλλον πω ότι διάφορες ε, χώρες έχουν νέα οικονομία ή αναδυόμενη οικονομία. Σε σχέση με τη χρήση όλων αυτών των πρακτικών, φαίνεται πως, ε, πως δεν υπάρχουν αρκούντως ε, ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Ακόμα πιο δύσκολο είναι για τις επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται σε απομακρυσμένες, ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές όπως οι Αζόρες ε, και η Μαδέρα. Τελευταία μου λέξη κύριε Πρόεδρε για τις αγορές εργασίας. Αναφέρω, καταρχήν πως δεν υπάρχουν δυνατότητες για συμβάσεις εργασίας, πράγμα το οποίο καθιστά δύσκολο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ορθολογικοποιήσουν τους ανθρώπινους πόρους τους και να αντιμετωπίσουν την κρίση. Το σύστημα το κοινωνικό δυσκολεύει περισσότερο τους επιχειρηματίες και καθιστά αυτή τη δραστηριότητα διόλου ελκυστική για την αντιμετώπιση της κρίσης. Πιστεύω από την άλλη πλευρά πως όλοι συμφωνούμε για το γεγονός ότι χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, όχι μόνο να περιορίσουμε όσο γίνεται περισσότερο ε, τον αντίκτυπο της κρίσης, αλλά να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο αυξημένης παραγωγικότητας. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για την εισαγωγική σας αυτή παρουσίαση. Θα περάσουμε στη Μαρία Νόβα τώρα και έγκαιρα ήρθε και ο τρίτος ημερογνώμα μας. Χαίρομαι που προφτάσατε. Σα χαιρετίζω καταρχήν η κυρία Νόβα και έχει το λόγο. Θα μιλήσω γαλλικά, αλλά η διαφάνιση είναι στα αγγλικά, για να τις παρακολουθείτε με μεγαλύτερη ευκολία. Θα σας μιλήσω κυρίως για την περίπτωση της Γαλλίας και τη γαλλική εμπειρία γέννη. Ναι, θα μιλήσω γαλλικά είπα, κυρίως για την κατάσταση στη Γαλλία, διότι στη Γαλλία έχουμε ε, μία ε, μη ε, τραπεζική οργάνωση από τις παλαιότερες που χορηγεί μικροπιστώσεις τα τελευταία 20 χρόνια 80.000 δάνεια έχει χορηγήσει έκτοτε σε ανέργους, σε άνθρωπους που ζουν με προνοιακά επιδόματα. Ε, 2,5% είναι οι απώλειες και 65% είναι η επιβίωση των επιχειρήσεων μετά από μια διετία που είναι και ο μέσος όρος στη Γαλλία γενικότερα. Χρειάστηκε και αλλαγή της νομοθεσίας και υποστήριξη ε, των τραπεζών που μας αναχρηματοδοτούν για τις πιστώσεις και στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης και του κράτους και της Ευρώπης βεβαίως για ε, τις συνοδευτικές ε, παροχές. Παρακαλώ την επόμενη διαφάνεια, θέλετε. Θα ήθελα λίγο να σας εξηγήσω το τοπίο των επιχειρήσεων στη Γαλλία, πώς διαγράφεται. 93% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες. Και στην Πορτογαλία περίπου το ίδιο συμβαίνει. Ε, και ε, προχώμε στην επόμενη διαφάνεια. στην Ευρώπη. Η κατάσταση είναι αντίστοιχη σε όλες τις χώρες. Δεν έχω όλα τα στοιχεία βέβαια για την Ευρώπη και ε, προτιμώ να παραμείνω στη Γαλλία. Αλλά η διάρθρωση και η δομή των επιχειρήσεων είναι αντίστοιχη σε όλη την Ευρώπη. Προχωρούμε στο επόμενο. Κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικό είναι να σας δείξω αυτές τις δύο καμπύλες των τάσεων Δυστυχώς δεν είναι πάρα πολύ καθαρή εικόνα και ευκρινής. Η ε, κόκκινη γραμμή που κατεβαίνει είναι ε, ο βιομηχανικός τομέας, ε, ενώ η πράσινη που έχει ενωδική πορεία είναι ο τριτογενής υπηρεσίες. Δηλαδή δείχνει ακριβώς μια βαριά τάση, έτσι μια πολύ μεγάλη τάση ε, προς την παροχή υπηρεσιών από πολύ μικρές επιχειρήσεις, από πολύ μικρές μονάδες. Γιατί σε αυτόν τον κλάδο φυσικά δεν χρειάζονται μεγάλα εργοστάσια, μεγάλα κεφάλαια, ούτε μεγάλο ανθρώπινο δυναμικό ως ε, υπάλληλοι. Η ίδια τάση ε, ενισχύεται από την άλλη από την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών τα νέα επαγγέλματα που αναδύονται για την προστασία του περιβάλλοντος, τη γύρα του πληθυσμού που βεβαίως ε, όλοι αυτοί οι παράγοντες ε, απαιτούν πλέον μια πολιτική απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας πιο ε, ενεργό. Και πάλι βλέπουμε ότι είναι μικρές οι μονάδες παραγωγής και οι μικροπιστώσεις λοιπόν ε, είναι το κατεξοχήν εργαλείο χρηματοδότησης σε μια πλέον μεταβιομηχανική εποχή της οικονομίας που διανύουμε. Πώς επηρέασε λοιπόν η κρίση την κατάσταση αυτή. Όπως βλέπετε ότι τα τελευταία 30 χρόνια εξελίχθηκε έτσι η κατάσταση. Στη Γαλλία το 2009 χάσαμε 500.000 θέσεις απασχόλησης. Και κατά την ίδια περίοδο δημιουργήθηκαν περίπου 600.000 νέες επιχειρήσεις. Δηλαδή, οι περισσότερες νέες θέσεις απασχόλησης προήλθαν από τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αξιοσημείωτο και αξιομνημόνευτο, στη Γαλλία αυτό ήταν μικρή επανάσταση. Ε, ε, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά η δημιουργία των επιχειρήσεων ε, αυξήθηκε κατά 72% και ε, για πολύ μικρές επιχειρήσεις το ποσοστό αυτό έφτασε στο 142%. Ο πρώτος σημαντικός λόγος είναι η κρίση. Βεβαίω, ο κόσμος από τη στιγμή που έχανε τη δουλειά του ως μισθωτό, ε, δημιουργούσε τη δική του θέση απασχόληση με μια προσωπική εταιρεία, ας πούμε. Και ε, φτάσαμε στους αυτοαπασχολούμενους. 300.000 ε, γράφησαν με το νέο καθεστώς αυτοαπασχολούμενοι από υπάλληλοι που ήταν πριν και έχαζαν τη δουλειά τους. Τώρα, 26.000 ε, είναι οι πελάτες ε, της ε, ΑΝΤΙ από πιο ευάλωτους κλάδους του πληθυσμού. Και είναι ιδιαίτερα ευάλωτες και έφραυστες αυτές οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και πλήγησαν ιδιαίτερα το μέσο του εισόδημα μειώθηκε και μειώθηκε πολύ κάτω από το κατόφλι της στόχιας, αλλά είναι αξιοσημωτή και πάλι ότι το 80% των πολύ μικρών επιχειρηματιών παραμένουν αισιόδοξοι, πράγμα που σήμερα είναι ιδιαίτερα σπάνιο και εξαιρετικό στον τομέα των επιχειρήσεων. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς τώρα. Η κρίση αυτή αποκάλυψε κάτι στη χώρα μας, αλλά δεν θα εκπλαγώ να ακούσω ότι συνέβη το ίδιο σε άλλες χώρες. γι' αυτό είναι ε, η ε, δημιουργικότητα που ε, τονώθηκε στη βάση της πυραμίδας. Και η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Ανάπτυξη των Μικροπιστώσεων υπέρ της ε, επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης ορίζει πάρα πολύ καλά το τι πρέπει να γίνει. Θα σας αναφέρω πολύ σύντομα τους τέσσερις άξονες της πρωτοβουλίας αυτής. Άξονας πρώτος ε, βελτίωση του νομικού και θεσμικού πλαισίου για τις μικροπιστώσεις, με σημαντικότερο εδώ σημείο κάποια ευελιξία στα επιτόκια, διότι οι μικροπιστώσεις απαιτούν για να καλύπτουν ε, το κόστος τους πιο ψηλά επιτόκια, τα οποία δεν βαρύνουν ιδιαίτερα ε, τους δανειστές, γιατί είναι μικρά δάνεια και για μικρή χρονική περίοδο και στη Γαλλία αλλάξαμε τον τραπεζικό νόμο και ε, καταφύγαμε στο δανεισμό εμείς από τις εμπορικές τράπεζες. Το επόμενο λοιπόν βήμα είναι να συνεννοηθούν οι δημοσιονομικές, οι χρηματοπιστωτικές αρχές των κρατών μελών για να βελτιωθεί αυτή η νομοθεσία. Ε, δεύτερος άξονας, ό,τι αφορά την νομοθεσία για τις μικρές επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους, και εδώ έγινε ε, μια βελτίωση και χρειάζονται βελτιώσεις και είναι η εξής. Χρειάζεται καλύτερη διάθρωση μεταξύ των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και δημιουργίας ε, της θέσης απασχόλησης ενός αυτοαπασχολούμενου. Και ε, κάποια πλαισίωση και βοήθεια για εκείνους που δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης και αυτοαπασχολούνται. Στη συνέχεια, τρίτος άξονας, ε, θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια ε, για μεγαλύτερη παροχή συμβούλων, εκπαίδευση, βοήθεια σε εκείνους που δημιουργούν την επιχείρησή τους. Η δράση αυτή τώρα ξεκινάει στο Jasmine που ε, ξέρετε ότι είναι ένα πρόγραμμα, μια πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης περιφερειακής ανάπτυξης όπου συμμετέχουν οι εταιρείε βαθμονόμηση οίκη ε, αυτή και τα ευρωπαϊκά δίκτυα. Και ο τέταρτος άξονας είναι να βρεθούν επιπλέον πόροι. Στην Ευρώπη είναι περιορισμένοι μάλλον και μεταξύ άλλων διότι το νομοθετικό πλαίσιο δεν τους επιτρέπει να είναι πιο ε, το 2008 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, επένδυσε 20 ε, δισεκατομμύρια ευρώ. 20 εκατομμύρια, συγγνώμη, και ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 4 εκατομμύρια και το 2010 ε, άλλα 3 θα προσθεθούν. Και το Δεκέμβριο 2009, όπως γνωρίζετε, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα μέσον 100 εκατομμυρίων για την επόμενη τετραετία. Συμπέρασμα. Η ανάπτυξη των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των μικροπιστώσεων ανταποκρίνεται πραγματικά στη νέα φάση της οικονομίας που διανύουμε αυτό τον καιρό. Έχουμε αποβιομηχάνηση παντού στην Ευρώπη. Δηλαδή, βεβαίως θα πρέπει να προσπαθήσουμε να σώσουμε ό,τι μπορούμε, αλλά να μην τρέφουμε και μεγάλες αυταπάτες. Βλέπουμε ότι 30 χρόνια μειώνεται ε, αυτή η τάση προχωρεί από βιομηχάνηση και δεν πρόκειται να αναστραφεί αυτή η πορεία. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να βγούμε από την κρίση. Δεν είναι ο μόνος, αλλά ένας από τους τρόπους. Στη Γαλλία λοιπόν χρειαστήκαμε 20 χρόνια για να βελτιώσουμε αυτό το περιβάλλον, το νομοθετικό και το θεσμικό. Γιατί χρειαστήκαμε 20 χρόνια, διότι στην αρχή ήμασταν στη Γαλλία ήμασταν τρει εθελοντέ και ήταν τελείω άγνωστη αυτή η προσπάθεια. Αλλά με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής νομίζω ότι στην Ευρώπη μπορεί να γίνει πιο γρήγορα αυτό και να έχει και απτά αποτελέσματα σε αυτούς τους τόσο δύσκολους καιρού. Η μεγαλύτερη δυσκολία τώρα δεν είναι να βρούμε κονδύλια γιατί βλέπετε ότι εμάς μας χρηματοδοτούν οι τράπεζες και δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα σε σχέση με αυτό. Εκτός, και αναλαμβάνω, από προσαρμογή του νόμου για τις τράπεζες, γιατί προηγουμένως οι τράπεζες δεν είχαν το δικαίωμα να μας αναχρηματοδοτούν. Άλλαξε ο νόμος όμως και κυρίως αυτό που χρειαζόμαστε τώρα για τις μικροπιστώσεις είναι κάποιοι ελάχιστη ήδη οι πόροι ή επιδοτήσεις για να καλύπτουν οι οργανισμοί αυτοί ε, το αρχικό τους κόστος μέχρι να μπει το νερό στα βλάκι και να έρχονται οι τόκοι και να ε, καλύπτουν τα έξοδά τους. Τώρα μπορούν και τα διορθωτικά ταμεία ε, πλέον να χρηματοδοτούν τις μικροπιστώσεις και την πλαισίωση και τη συνοδεία τους, αλλά σήμερα τα διορθωτικά ταμεία δεν επιτρέπουν να κρατάμε τους τόκους και να σταθεροποιούμε κάπως το σύστημα και να το κάνουμε αηφόρο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Από την Πορτογαλία πήγαμε στη Γαλλία, τώρα περνάμε στην, στο βορρά της Ευρώπης. Έχουμε τον κύριο Πράουνχελμ. Δέκα λεπτά να μας κάνει μια παρουσίαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλη μου ευχαρίστηση που είμαι εδώ. Εγώ θα κάνω μια σύντομη παρουσία της υποδομής, να πω δύο λόγια τι μπορούμε να περιμένουμε και μετά κάποια συμπεράσματα όσον αφορά την πολιτική που πρέπει να ακολουθεί. Τι διαβλέπουμε τώρα. Είναι πια έντονη ολοκλήρωση παλιών και νέων χωρών στην παγκόσμια οικονομία. Αυτό σημαίνει ότι ενδυναμώνεται ο ανταγωνισμό. Ταυτόχρονα όμω βλέπουμε να υπάρχει ένα ανταγωνισμό μεταξύ των ήδη βιομηχανικών χωρών. Όσε μελέτε γίνονται, καταδεικνύουν ότι περίπου 50% των, της παραγωγής θα περάσει στις πιο ε, πρόσφατα ο βιομηχανικές χώρες, ως, τουλάχιστον όσον αφορά την απαραγωγή που δεν βασίζεται σε πάρα πολλές γνώσεις. Θα, όσον αφορά το παγκόσμιο εργοδοτικό δυναμικό, αντιμετώπισε έντονο ανταγωνισμό από το 2009-2025 υποθέτει ότι θα αυξηθεί και ακόμη περισσότερο το 2025-2030. Η γνώση είναι σημαντικό συστατικό για να προωθηθεί η ανάπτυξη. Οι γνώσεις αυτές θα πρέπει βέβαια να μετατραπούν σε μια οικονομικά βιώσιμη γνώση. Αυτό σημαίνει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που δίνουν τη δυνατότητα να ε, συλλέξουμε στοιχεία ότι αυτό έτσι πραγματικά συμβαίνει. Αυτό που είναι επίσης σημαντικό για την καινοτομία είναι ε, ότι υπάρχουν συχνά πολύ ριζοσπαστικές καινοτομίες που οδηγούν και σε ανάπτυξη της απασχόλησης. Θα σας δείξω κάποιες διαφάνειες που να παρουσιάσουν αυτή την κατάσταση από την ε, έκθεση της ε, Σουηδικής, ε, του Σουηδικού αυτού Συμβουλίου. Βλέπετε εδώ έχουμε μια κατανομή της παραγωγής ανάλογα κατά πόσον βασίζεται στις γνώσεις ή στο κεφάλαιο ή στις ικανότητες των εργαζομένων. Και βλέπετε τις διαφορές που υπάρχουν και τα επόμενα 4-5 χρόνια θα υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερες διαφορές. Ανάλογα κατά πόσον η παραγωγή βασίζεται σε κεφάλαιο, σε γνώσεις ή στο εργατικό δυναμικό. Τα πράγματα δεν είναι πολύ εύκολα βέβαια, αλλά υπάρχουν πολύ έντονε προσδοκίε για τη μικρομεσαία επιχειρήση στον τομέα που βασίζεται ακριβώ στι γνώσει. Αν κοιτάξετε την άλλη διαφάνεια, βλέπετε ότι η μπλε αυτή ε, καμπύλη αναφέρεται στην ε, επιστροφή σε πιο εκπαιδευμένο προσωπικό, ενώ η άλλη κάτω η κόκκινη που κατεβαίνει ε, αποδεικνύει τους του ποια είναι τα ε, έσοδα των λιγότερο εκπαιδευμένων εργαζομένων. Αυτές οι αλλαγές οδηγούν σε σημαντικές προκλήσεις τους πολιτικούς. Άμα δούμε από πού ξεκίνησε η απασχόληση. Στην πρώτη γραφική παρουσίαση, στα αριστερά σας δηλαδή, βλέπουμε τις 30 μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην Σουηδία και η απασχόληση, ανάλογα αν η απασχόληση αυτή είναι στο ιστορικό της χώρας ή στο εξωτερικό. 75 2005 δεν υπήρχε μεγάλη διαφορά, αλλά όπως βλέπετε στο σκοτεινό τμήμα, μειώθηκε σημαντικά το ποσοστό αυτό της απασχόλησης στη Σουηδία, μέσα την ίδια, και αυτό είναι απαραίτητο για να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι η απασχόληση αυξήθηκε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στον παραγωγικό τομέα. Ιδίω ακόμη περισσότερο στον τομέα των υπηρεσιών χαμηλού επίπεδου. Εδώ βλέπετε την κατανομή στον τομέα του υψηλού, της υψηλής ε, προσφοράς ε, υπηρεσιών. Όπου βλέπετε ότι υπάρχουν πραγματικά μετατροπές και μια τάση προς περισσότερη απασχόληση στο δομέα των υπηρεσιών. Ποιες είναι οι ιδέες των ΜΜΕ και πώς έχουν πληγεί από τις κρίσεις. Αυτή η διαφάνεια σας δείχνει πώς ε, αντιμετωπίζουν τις ε, επιρρησιακές ευκαιρίες. Ε, ανάλογα κατά πόσο πρόκειται για καινούριε παλιές ε, Εταιρείε ή εταιρείες οι οποίες συνεχίζουν να δρούν και βλέπετε τι γίνεται. Θα πρέπει να δείτε το, τη γαλάζια στήλη εκάστοτε που αναφέρει τις οικονομίες που βασίζονται στην καινοτομία και εκεί βρίσκονται οι περισσότερες ε, χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε αυτό το τομέα. Αυτή η διαφάνεια βασίζεται σε διάφορες ε, πηγές ε, στοιχείων, αλλά όλες οι πηγές οδηγούν στα ίδια αποτελέσματα. Σημαντική μείωση των ευκαιριών, όπως λαμβάνω υπόψη, και όσον αφορά την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, έχουμε χαμηλή παρουσία των λεγόμενων λαφιών, γκαζέλ. Χαμηλές προσδοκίες από εκείνους που έχουν την ψηλότερη εκπαίδευση. Είναι πάρα πολύ αρνητικό αυτό αύξηση στον φόβο αποτυχίας και αύξηση στην ε, επιμαστική δράση που βασίζεται στις αναγκαιότητες. Σα είπα υπάρχει επίση παρόμοια εικόνα. Το 85% θεωρούν ότι είναι κακή εποχή αυτή να ξεκινήσουμε επιχείρηση. Το 65% λένε ότι υπάρχει μείωση του κύκλου εργασιών και της αποδοτικότητας και το 1 τρίτο έχουν μειώσει τον αριθμό των απασχολουμένων. Και η έλλειψη διαθεσίμων κεφαλαίων για δανειοδότηση έχει πλήξει περισσότερο τις ΜΜΕ, οι οποίες έχουν μειώσει σημαντικά κατά ένα τρίτο μάλιστα τις ε, δαπάνες για την έρευνα και την ανάπτυξη. Και αυτό είναι σημαντικό βέβαια για να εξασφαλίσουν τη μελλοντική τους ανταγωνιστικότητα από την άλλη μεριά. Τι μπορεί να γίνει τώρα. Έλλειψη ζήτηση. Και η Μακροπολίτη έκανε ό,τι μπορούσε. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά στο επίπεδο των μακροοικονομικών πολιτικών. Εδώ έχουμε μία διαφάνεια η οποία δείχνει τη σχέση μεταξύ την προστασία της αγοράς απασχόλησης και τις προσδικίες μικρομεσαίων επιχειρήσεων όσον αφορά τις μελλοντικέ τους προσδικές ανάπτυξης και βλέπετε ότι η σχέση είναι αυστηρά αρνητική. Δεν λέει η διαφάνεια αυτή γιατί, πάντως η σχέση είναι αρνητική. Τώρα, επίσης, οι φόροι ε, Corporate seems to be... Uh, είναι το πιο σημαντικό. Οι, οι φόροι για τις ε, επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας στην ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης. Και βλέπετε ότι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν σημαντικά επίπεδα ε, επίπεδα φορολογικής επιβάρυνσης. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οι πολιτικές να καλύπτουν πάρα πολλούς τομείς. Δεν μπορούμε να εξετάσουμε μόνο την αγορά απασχόλησης Φερρυπίν. Θα πρέπει να καλύψουμε περισσότερα από τις μακροοικονομικές πτυχές και πιστεύω ότι τέσσερις είναι σημαντικές. Γνώσεις, αγορά απασχόλησης, καινοτομία και δυνατότητα ανανεωση μια επιχειρήση και φόρου. Θα σας πω δύο λόγια για κάθε έναν από τους τομείς αυτούς. Ε, αυξήθηκε σημαντικά η κρατική έρευνα και ανάπτυξη, αλλά μπορούν ακόμη πολλά να γίνουν να αυξηθεί. Εκτός αυτού θα πρέπει να φροντίσουμε, να προσελκύσουμε και να διατηρήσουμε εκείνες τις μεγάλες εταιρείες που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι πάρα πολύ σημαντικοί επενδυτές στην έρευνα και την ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε περισσότερη επιχειρησιακή δραστηριότητα που να βασίσει στην τεχνολογία. Και θα πρέπει εδώ να δούμε τα λεγόμενα voucher για την έρευνα και ανάπτυξη, να προωθήσουμε την σχέση μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστημίων ή ερευνητικών κέντρων. Θα πρέπει να προσελκύσουμε ταλέντο θα πρέπει λοιπόν να είμαστε εξή ελκυστικοί όσο άλλε χώρε. Αγορά απασχόληση, να δημιουργήσουμε προποθέσει που οδηγούν σε διαθετικέ αλλαγέ. Χρειαζόμαστε ευελιξία, χρειαζόμαστε ισχυρά ιδρύματα εκπαίδευση και ε, μετεκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση. Θα πρέπει ίσω να αλλάξουν κάποιε δομέ εκεί. Μετά, οι, εξ, αποταμιεύσεις για τη σύνταξη θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους εργαζόμενους για τη δική τους εκπαίδευση, αν θέλουν. Υπάρχουν κάποια σφάλματα και ο τίτλος του θα πρέπει να είναι ε, όχι SMEs και entrepreneurship, αλλά ε, καινοτομία και δυνατότητα ανανέωσης οι πολιτικές εξόδου, ε, πτώχευση, τα κίνητρα για κεφάλαιο κινδύνου, πολλές δυνατότητες ε, βελτίωσης στα θεσμικά όργανα. Ο ανταγωνισμός θα πρέπει να ενδυναμωθεί. Ο δημόσιος τομέας εξακολουθεί να έχει ένα μεγάλο ποσοστό, ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών. υπάρχει και πάρα πολύ ενίσχυση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στη χώρα μου, παραδείγματος χάρη, πολύ λίγες δυνατότητες δίνονται για την γνώση της αγοράς, παγκοσμιοποίηση κλπ. Και θα πρέπει η υποστήριξη να κατευθύνεται προς την κατεύθυνση αυτή μέσα στα πλαίσια βέβαια του τι υπάρχει αυτή τη στιγμή. Οι φόροι αναφόρθηκαν ήδη, η ισορροπία μεταξύ των προσωπικών ε, φόρων και των φόρων κεφαλαίου, η διαφάνεια, η ομοιομορφία των φορολογικών συστημάτων. Επίσης, η στάση, οι παραδόσεις, ε, τα πρότυπα είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρος, εγώ σας ευχαριστώ. Περνάμε στα ερωτήματα τώρα. Μία, α, δύο ερωτήσεις. Ναι. Έχουμε κάποιες εδώ. Θα αρχίσουμε με το ΕΛΚ και θα περάσουμε στους ε, σοσιαλδημοκράτες, Πράσινε, Πράσινες, εγώ και αυτά. ΕΛΚ, Πάστος και ΦΕΟ. Muito obrigada, Sr. Presidente. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές που παρενέβησαν στο πρώτο τμήμα αυτής της ακρόσης και σαφώς ε, να τους ευχαριστήσω γιατί μας εξέθεσαν τις εθνικές τους εμπειρίες σε σχέση με τον αντίκτυπο της κρίσης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εγώ θα ήθελα να απευθύνω μια ερώτηση στον συμπατριώτη μου, τον ε, δόκτορα Αντώνιο Σαράιβα, πρόεδρο της, ε, του Πορτογαλικού ΣΕΒ. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξή, ε, κυρία Σαράιβα. Εμεί γνωρίζουμε ότι στην Πορτογαλία οι μικρομεσαίε επιχειρήσει ε, είχαν ένα επιπλέον πρόβλημα το οποίο επιδεινώθηκε με την κρίση και επίσης έχουν ιδιαίτερα προβλήματα που σχετίζονται με το την εθνική τους πλαισίωση. Έχει να κάνει με την επιλογή της πορτογαλικής κυβέρνησης υπέρ των μεγάλων δημοσίων έργων, τις επενδύσεις υπέρ των μεγάλων δημοσίων έργων εις βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά έχουμε επίσης μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση των πληρωμών από πλευρά του προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πράγμα οποίο δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες στις τόσο αυτές σημαντικές δομές διατήρησης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Και έχουμε ένα πολύ ιδιαίτερο επίσης πρόβλημα που έχει να κάνει με το δικαστικό σύστημα, την πολύ δυσκίνητη μηχανή του και την ε, καθυστέρηση στην επιβολή των ε, αποφάσεων. Ε, θέλω Θέλω λοιπόν να γνωρίζω ότι έχουμε προβλήματα στην Πορτογαλία τόσο όσον αφορά τις πιστώσεις, όσον αφορά την ε, φορολογία, όσο, τόσο όσον αφορά τον έλεγχο. Ποια είναι τα μέτρα που εσείς ε, θα βλέπατε για να μπορέσετε να απαντήσετε σε αυτό το θέμα για τους άλλους ομιλητές. Θα ήθελα να γνωρίζω επίσης αν στις δικές σας χώρες υπήρχε πραγματικά συγκέντρωση των ε, παραγόντων που επηρεάζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε κάθε χώρα ποιοι ήταν αυτοί οι παράγοντες οι οποίοι επιδεινώθηκαν περισσότερο μέσω της χρηματοοικονομικής κρίσης. Ευχαριστώ. <clears throat> σε σχέση με την ε, ερώτησή σας, με το ότι, γεγονός ότι η κυβέρνηση ευνοεί τα δημόσια έργα ε, και καθυστερεί τις πληρωμές σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να σας πω, η δική μας άποψη είναι ότι δίνοντας ε, πόρους σε δημόσια έργα, αυτό σημαίνει πως υπάρχουν χρήματα Και εφόσον αυτά τα χρήματα υπάρχουν για τα μεγάλα δημόσια έργα, για το ΤΖΒ, το αεροδρόμιο, βλέπουν ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να περιορίζονται ε, χωρίς να μπορούν να πάρουν ένα μερίδιο από τα κονδύλια αυτά ή, πάση περιπτώσει, με το να περιορίζονται σε ψίχουλα. τα δημόσια έργα θα πρέπει βασικά να βλέπουν την παρέμβαση του πορτογαλικού επιχειρηματικού κόσμου, ώστε στην κατανομή των ε, έργων σε μια πολιτική εγκύτητας να μην δίνονται πόροι μόνο για τα μεγάλα αυτά έργα που άμεσα θα γίνουν. Θα πρέπει δηλαδή να εξισορροπηθούν όλα αυτά γιατί αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτές οι οποίες δημιουργούν τις θέσεις απασχόλησης. Μόνο 800 μεγάλες επιχειρήσεις υπάρχουν στην Πορτογαλία. Θα πρέπει λοιπόν υπάρξει μια διαφορετική εθνική πολιτική ώστε το, η πίτα αυτή που κάθε τόσο μικραίνει να μοιραστεί πιο δίκαια και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να σας πω κάτι που την ημέρα που ανέλαβα τα καθήκοντα αυτά ε, είπα θεώρησε ότι η δικαιοσύνη θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματική, πιο ταχύρυθμη, γιατί με την καταβολή των πληρωμών που, ανέ, που σας ανέφερα, στην, πράγματι η Πορτο, στην Πορτογαλία υπάρχει αυτή η χείριστη πρακτική, δηλαδή να καθυστερούν τις πληρωμές όλοι όσο γίνεται περισσότερο, ακόμα και σε 2.000 μέρες καθυστέρηση, δηλαδή μιλάμε για καθυστέρηση 4-5 ετών στην καταβολή των ε, πληρωμών. Αυτή λοιπόν η χαλαρότητα στις πληρωμές και η δικαιοσύνη η οποία δεν βοηθά, σέρνονται οι υποθέσεις για χρόνια και χρόνια στα δικαστήρια χωρίς να βγαίνει απόφαση και χωρίς να, ε, να, να βοηθούνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή χάνουν τις, ε, τις, ε, ε, παραγγελίες, δεν θα έχουν κέρδη, είναι υποχρεωμένοι να δώσουν μια πληρωμή για κέρδη τα οποία δεν θα πάρουν και συνέχεια αυξάνεται αυτή και αυξάνονται διαρκώς οι δυσκολίες που υπάρχουν. Χρειάζεται λοιπόν καλύτερη πολιτική όσον αφορά τον έλεγχο. Πρέπει να εξελιχθούμε Δεν, δεν γίνεται διαρκώς να αλλάζει το φορολογικό πλαίσιο το οποίο τιμωρεί και αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Κυρία Νοβάκ, εγώ πιστεύω ότι όπως παντού και στη Γαλλία οι μικρομεσαίες είχαν ένα πρόβλημα ζήτησης. Και αυτές που συνδέονται με την ε, αυτοκινητοβιομηχανία, τις βιομηχανίες που είχαν δυσκολίες, είναι αυτές οι οποίες υπέφεραν και περισσότερο. Αυτά που έγιναν από την κυβέρνηση ήταν ε, βασικά να δώσουν στις τράπεζες πιστώσεις που επέτρεπαν να αυξήσουν τα δάνεια. Και επιπλέον ένας διαμεσολαβητής για τις μικρομεσαίες που δεν κατάφερναν να πετύχουν δάνεια. Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει δύσκολη, όπως παντού. Sorry, uh, I think that, uh... Συγγνώμη. Ε, πολλά από αυτά που είπατε ισχύουν και για τη δική μου χώρα και για πολλές ακόμα. Πολύ συχνά είναι πολύ μεγάλη η γραφειοκρατία, δεν χωράει καμία εμφιβολία και το νομικό σύστημα είναι εξαιρετικά αργό. Όταν μιλάμε για εκπρόθεσμη ε, πληρωμή τιμολογίων, εκεί δεν ενέχονται μόνο δημόσιοι φορείς, αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις το χρησιμοποιούν αυτό. Και αυτό είναι ανάρμοστο για μένα. Και οι κανόνες επίσης για τις ε, προμήθειες του δημοσίου και τα δημόσια έργα είναι δύσκολοι στη χρήση του, στην ε, εφαρμογή τους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Χρειάζεται λοιπόν ένα καλό νομικό και θεσμικό πλαίσιο για να έχουν ευκαιρίες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για τα δημόσια έργα βέβαια αυτό είναι περιορισμένο και σε χρονική διάρκεια και σε αντικείμενο. Δεν μπορεί κανείς να το έχει ως πάγια ε, μακροχρόνια στρατηγική. Και σταματώ εδώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε. Αναδύω τώρα οι ερωτήσεις και παρακαλώ να επικεντρώσετε στις ερωτήσεις, μην κάνετε σχόλια. Και η δυνατό ε, ένα-ενάμιση λεπτό, γιατί είστε πολύ απίθαρχοι. Ο κύριος Φέο και μετά ο κύριος Κάρας. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές που είχαμε απόψε. μιλήσατε για την ανάγκη ευελιξίας ε, της ε, αγοράς εργασίας. Ε, ήθελα να σας ευχαριστήσω γι' αυτό και η αναφορά που μας κάνατε όσον αφορά την απλοποίηση των κανόνων. Εγώ θέλω μια ερώτηση να απευθύνω και στους τρεις σας. Ένα από τα θέματα που ήταν κοινό σε όλες τις παρεμβάσεις ήταν η πίστοση και η σημασία της πίστοσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε μια περίοδο που ήδη αρχίζουμε να ακούμε για στρατηγικές ε, διαφορετικό βέβαια σύστημα σε κάθε κράτος και δεκούμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν μεγάλες δυσκολίες ε, να πάρουν πιστώσεις για να μπορέσουν να επενδύσουν. Θα ήθελα να ξέρω τι ρόλο πιστεύετε πως μπορεί να παίξει το κράτος ή, εν πάση περιπτώσει, οι μονάδες ε, δημόσιου χαρακτήρα όπως ας πούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με αυτό το θέμα. Δηλαδή, πώς μπορούν να στηρίξουν το οικονομικό σύστημα ώστε να μπορέσουν να στηρίξουν την προϋπόθεση των πιστώσεων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε ποιον απευθύνεται την ερώτηση. Ότμα. Ότμαρ Κάρας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ για τις τοποθετήσεις σας. Έχω δύο ερωτήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια νομοθεσία πρότεινε για τις μικρές επιχειρήσεις, Small Business Act. Εμείς έχουμε λίγες αρμοδιότητες για να το επιβάλλουμε αυτό στα κράτη-μέλη. Ποιες ευκαιρίες βλέπετε εκεί, πιο δυναμικό θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε εάν υλοποιηθεί 100% αυτό το πρόγραμμα στα κράτη-μέλη και τι πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε να προωθήσουμε και, ε, την αρχή αυτή small business first, πρώτα οι μικρές επιχειρήσεις. Ποια είναι τα βασικά εμπόδια και εσείς τι ε, απαιτήσει έχετε από την Ευρώπη του 2020. Τι θα πρέπει να ορίζει αυτό το πρόγραμμα για το 2020 για να γίνουν όλα αυτά πραγματικότητα. Σε ποιο, ποιο ρωτάτε ε, βασικά τους δύο πρώτους ομιλητές. Oui, je, je suis pas sûr de, de pouvoir répondre. Δεν είμαι βεβαία ότι μπορώ να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Αυτό μπορώ να πω σε σχέση με την πρώτη ερώτηση είναι ζητάμε από το κράτος κάτι πολύ δύσκολο γιατί από τη μια πλευρά θέλουμε να, να δώσει όθεση να στηρίξει τις πιστώσεις αλλά από την άλλη πλευρά να αποφύγει την ε, υπερχρέωση. Άμα ο δανεισμός είναι δύσκολος, αυτό οφείλεται επίσης γιατί η οικονομική κατάσταση είναι δύσκολη και ε, επειδή στο ότι η ζήτηση είναι μικρή. Αντικειμενικά λοιπόν πιστεύω πως δεν είναι και τόσο εύκολο αυτό. Και το βλέπω και σε επίπεδο των πελατών μας, όπου δεδομένης αυτής της αδυναμίας, της, της μικρής μάλλον πρέπει να προσέχουμε περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, να μην υπερχρεωθούν οι άνθρωποι που θέλουν να αναπτύξουν την εταιρεία τους, την επιχείρησή τους. Τώρα, για εκείνο την νομοθεσία για τις μικρομεσαίες δεν μπορώ να σας δώσω πλήρη απάντηση. Εγώ νομίζω πως όλα όσα κατευθύνονται προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι εξαιρετικά σημαντικά, διότι είδατε και παρουσιάστηκε και στην περίπτωση και των τριών χωρών πως αντίθετα από αυτό που πιστεύουμε δεν είμαστε πλέον μια μεγάλη βιομηχανική οικονομία ή περισσότερες εταιρείες στην Ευρώπη είναι μικρές, πολύ μικρές. Και ό,τι άρα μπορεί να ευνοήσει τη δημιουργία και την ανάπτυξη αυτών των μικρών επιχειρήσεων, θα οδηγήσει στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Thank you. Uh, I think one of the fundamental... Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι ένα από τα βασικά προβλήματα είναι ότι ε, στην Ευρώπη χρηματοδοτούμε ε, πολύ τα δάνεια ε, και αλλά χρειαζόμαστε περισσότερες μετοχές, δηλαδή ίδιο κεφάλαιο ιδιώτες επενδυτές και όχι επιδότηση και χρηματοδότηση δανείων ε, συμπληρωματικά με τα όσα συμβαίνουν ε, τώρα. Βεβαίως θα μπορούσαν να επεμβαίνουν οι κυβερνήσεις ε, όταν έχουμε τέτοιες κρίσεις για περιορισμένο χρόνο με συγκεκριμένες εγγύησεις, όπως έκαναν άλλωστε και τα κράτη. Και έτσι μπόρεσαν να δοθούν δάνεια για εξαγωγές και τέτοια Πάντως, όταν αποτυγχάνει η αγορά θα πρέπει να είναι παρούσα η κυβέρνηση, αλλά δεν είναι καλή ιδέα να επιδοτούμε μονίμως και συνεχώς ε, ε, δάνεια ε, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Καλύτερα είναι να δημιουργηθούν θεσμοί ιδιωτικοί που να αναλάβουν αυτή την ευθύνη και όχι το κράτος. Ευχαριστώ. Ε, σε σχέση με τις επιστώσει, εγώ αναγνωρίζω ότι θα πρέπει να υπάρξουν κατά τη διάρκεια τουλάχιστον αυτού του έτους, του 2010, αυτές οι ε, ε, η πορτογαλική κυβέρνηση το στηρίζει αυτό. Εμείς πιστεύουμε πως όλα αυτά έχουν μοιραστεί λάθος. Δεν σημαίνει βέβαια πως δίνοντας χρήματα θα λυθούν τα προβλήματα. Ήδη έγινε μια σχετική ανάλυση. Οι επιχειρήσεις που δεν προσαρμόστηκαν δεν θα επιβιώσουν και στην ουσία γίνεται στρέβλωση της κατάστασης. Δεν είναι υγιής αυτός ο ανταγωνισμός και είναι μια πρακτική την οποία δεν επιθυμούμε. Κάθε εταιρεία είναι μια συγκεκριμένη περίπτωση, κάθε τομέα δραστηριότητα είναι ξεχωριστό. Θα πρέπει τα χρήματα να κατευθυνθούν σωστά, να δρομολογηθούν σωστά και να βοηθηθούν εκείνοι που έχουν τη δυνατότητα να μετατροπεί σε μεταρρύθμιση προσαρμογή στον νέο κόσμο, στη νέα πραγματικότητα που δίνει όθηση σε πιο προηγμένα τεχνολογικά προϊόντα και όπως σας είπα και στην αρχή δεν είναι ρίχνοντας χρήμα ότι θα λυθούν τα προβλήματα. Θα πρέπει λοιπόν να βοηθηθούν όλοι, αλλά με, το, ένα ισόρροπο τρόπο. Τώρα για την σχετική νομοθεσία της Κομισιόν, ό,τι υπάρχει για να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ευπρόσδεκτο. Ευχαριστώ. Κλείνει ο κατάλογος. Οκτώ ακόμα υπερβάνς και μετά Κοφεράτη. Όλε Σμιτ από τους φιλελευθέρους και Σβίμπερ ε, από τους συντηρητικούς και μετά πάλι συντηρητικοί, Κάριντς, σοσιαλιστές, Γιακόν Σάρη και εγώ τελευταίος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να υπάρξει Small Business Act. Διότι πιστεύω ότι είναι σημαντική για μας τους νομοθέτες εδώ η ερώτηση του Ότμαρ Κάρας για σας και αυτή την ερώτηση απευθύνω και στους τρεις. Μέχρι ποιο σημείο θεωρείτε ότι πρέπει να ενισχυθεί αυτό το μέσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πρόσβαση των μικρομεσαίων είναι κρίσιμο θέμα ε, θέματα των δημοσίων έργων. Και η δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με το εξής διακύβευμα. Με ποιον τρόπο οι μικρομεσαίες, γιατί μικρομεσές, οι εντάξει όλες οι μικρομεσαίες, ε, υπάρχουν και πάρα πολλοί μικρές που κανονικά δεν εντάσσονται και αυτό είναι σφάλμα. Γιατί αποκλείονται και από κάποια χρηματοδότηση. Λοιπόν, αυτός ο κλάδος πώς ε, αντέδρασε από πλευράς κοινωνικού αντικτύπου της κρίσης. Δηλαδή, σε σχέση με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, πώς μπόρεσε να απορροφήσει αυτό το κοινωνικό κραδασμό. Γιατί έχουμε την εντύπωση ότι οι μικρομεσές ε, διατήρησαν το δυναμικό τους το ανθρώπινο. Γιατί υπάρχει κίνδυνο κάποιοι εργαζόμενοι που εκπαιδεύτηκαν στην επιχείρηση και κάποια στιγμή όταν σφίγγουν τα πράγματα φεύγουν από την εταιρεία, δεν μπορούν να ανακτηθούν όταν ε, ανακάμπτει η οικονομία. Λοιπόν, απορρόφησαν αυτούς τους κοινωνικούς κραδασμούς οι μικρομεσαίες ή απέλησαν Σε ποιον απευθύνει την ερώτηση του, σου την πρώτη και στους τρεις, στη δεύτερη. Στη δεύτερη όποιος θέλει. Εσύ αποφασίζεις. Κοφεράτη. La domanda è rivolta... Ο Η ερώτησή μου είναι για τον ε, Δόκτωρο Σαράιβα και τον Δόκτωρο Μπράουνερ Λέιν. Στη γλώσσα μου είναι δύσκολο το όνομά σας να το προφέρω, με ζητώ συγγνώμη. Το ερώτημα είναι το εξής. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα όπου η μικρή επιχείρηση ιστορικά αποτελούσε ένα στοιχείο ευελιξίας ε, του οικονομικού παραγωγικού συστήματος. Πάρα πολλές φορές, ε, κατά τη διάρκεια των αρνητικών κύκλων που χτυπούσαν ε, τις μεγάλες επιχειρήσεις, η μικρή αντιστάθμιζε το πλήγμα. Αυτή τη φορά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οι δυσκολίες στις μικρομεσαίες στάσαν αργότερα, αλλά με μεγάλη ένταση. Νομίζω λοιπόν ότι ήδη θα πρέπει να γίνει μια πρώτη διάκριση ανάμεσα στη μικρή επιχείρηση που έχει ένα προϊόν με ψηλή προστάμενη αξία και τη μικρή βιοτεχνία. Δεν αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο. Και ακριβώς ε, το μόνο σημείο που τις ενώνει είναι η δυσκολία πρόσβαση στις πιστώσεις, το οποίο αναφερθήκατε κι εσεί. Αλλά πέρα από τη σχέση με τι κυβερνήσει. εγώ θα ήθελα να γνωρίζω αν κατά την άποψή σα χρησιμεύει σε οτιδήποτε, σε κάτι, εν περιπτώσει, η δημιουργία σχέσεων ανάμεσα σε αυτές τι επιχειρήσει. Δηλαδή, αν οι μικρομεσαίε επιχειρήσει που βρίσκονται στην ίδια περιοχή, ακόμα και σε σχέση με τις διοικήσει που έχουν πολιτικέ που είναι διαθέσιμες για να προωθήσουν την ανάπτυξη των μικρομεσαίων, αν θα ήταν καλό, χρήσιμο, να τις οθήσουμε να ε, συνεργαστούν, να δημιουργήσουν δηλαδή μια κρίσιμη μάζα όσον αφορά τα στοιχεία που αφορούν την έρευνα και την γνώση. Oui. Euh, euh, Écoutez, je, je voudrais peut-être commencer par, par la première question. Για να απαντήσω, ναι, σε μια περίοδο κρίσης θα πρέπει ακριβώ να δημιουργηθούν δίκτυα για να ενδυναμωθεί να, ε, η δομή αυτή των ΜΜΕ και μέσα στα πλαίσια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το έχω ήδη δει στο παρελθόν και βλέπω και μέσα στα πλαίσια του ε, ευάλωτου πολίτη που έχουμε μπροστά μας και θα πρέπει να υπάρξουν κάποια συστήματα που θα επιτρέπουν αλληλέγγυα να προωθηθεί μια τέτοια δικτύωση στον τομέα των, ε, της έρευνας και της ανάπτυξης και μετά να προωθούν ε, τα ίδια θέματα με οτιδήποτε τρόπο θα ήταν ο ιδανικός. Νομίζω ότι έτσι μπορούμε να καλύψουμε όλες ε, τις ε, συνελτηριστικές εμπειρίες του 19ου αιώνα. Σχετικά δε με το ερώτημα της κυρίας Περές. για το Small Business Act είναι σημαντικό νομίζω. να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις δημοσιογορές. Και στη Γαλλία οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έπαιξαν ένα ρόλο κοινωνικού αμορτισέρα γιατί ακριβώς ε, δεν υπέστησαν ίσως τόσο πολύ τα διάφορα σοκ. όπως κάποιες άλλες βιομηχανίες. Απέλησαν βέβαια και οι ΜΜΕ. Δεν μπορώ να σας απαντήσω λοιπόν με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Κατ' εμένα όμως πραγματικά αυτό αυτός ο συστός των μικροεπιχειρήσεων και των ΜΜΕ λίγο πιο μεγάλων είναι η βάση της οικονομίας σας που συμπεριλαμβάνει ένα σχετικό μικρό αριθμό μεγάλων επιχειρήσεων που υποφέρουν περισσότερο βέβαια και από την κρίση η ερώτηση που θέσατε και κύριε Κομφεράτη, ναι, δεν απορροφούν τα εργατικά χέρια που έμειναν χωρί δουλειά, γιατί και αυτές οι ίδιε βρίσκονται σε φοβερή κατάσταση. Δεν έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν ε, τα προγράμματά σα, δεν μπορούν ε, να σταθούν. Τα ίδια τα κεφάλαια των εταιριών ε, είναι λιγοστά, είναι σε μια κατάσταση που τελικά οδηγεί και αυτές τις μικρομεσαίες να απολύουν. Γι' αυτό και αυξάνεται τόσο η ανεργία σε σχέση με την ερώτηση του κ. Κομφεράτη για την συνεργασία μεταξύ των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι κατά την άποψή μου ο μόνος δρόμος. Εμείς έχουμε φτιάξει μία οργάνωση, εγώ κατασκευάζω ας πούμε βρύσες και προσπαθούμε να φτιάξουμε κλάδος, κλαδικές ας πούμε και πρέπει αυτό να επεκταθεί σε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αν σκεφτεί κανείς ότι ε, έχει ας πούμε να φτιάξει κάποιο ένα μπάνιο και εσύ πας και του προσφέρεις μόνο τη βρύση, δεν θα προτιμήσει εσένα θα προτιμήσει τον άλλον που θα έρθει με την πανιέρα, το νεροχύτη, την ε, τουαλέτα, τις βρύσεις και όλα. Ε, για, είναι πολύ σημαντικό να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε αυτή την πιο δύσκολη αγορά. Μαζί, σίγουρα, ενωμένοι, θα είμαστε πιο ικανοί να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις ναι, όπως ελέγχθηκε προηγουμένως, πιστεύω ότι το Small Business Act, ο νόμος για τις μικρές επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ σημαντική. Οι πολιτικές για την αγορά απασχόλησης είναι επίσης πάρα πολύ κρίσιμες, γιατί εκείνες θα εξασφαλίσουν ότι η οικονομία δεν θα βρεθεί να αντιμετωπίζει ένα τεράστιο αριθμό απολυμμένων εργαζομένων. Υπάρχουν βέβαια διαφορετικές πρακτικές μεταξύ των χωρών και μπορούμε να μάθουμε από τις καλύτερες πρακτικές βέβαια. Τώρα συνεργασία φυσικά πάρα πολύ σημαντικό. Μικρές επιχειρήσεις, μικροεπιχειρήσεις χρειάζονται οπωσδήποτε να διαβεβαιωθούν ότι εισακούεται η φωνή τους. Και αυτό δημιουργεί μια κουλτούρα αν θέλετε περιφερειακής αλληλεγγύης. Και ξέρετε σε χώρες που υπάρχουν οι παρόμοιες ε, πρακτικές, υπάρχουν παρόμοιες προϋποθέσεις, υπάρχουν διαφορές λόγω των διαφορετικών πρακτικών. Και θα ήταν καλό να υπάρχουν νέα δίκτυα. Ευχαριστώ, πρόεδρος. Ευχαριστώ. Έξι έχουν ακόμα φαλερωτήσεις. Ε, ε, τρεις και τρεις θέλουμε, γιατί δεν θέλω να χάσουμε από το δεύτερο πάνελ το χρόνο. Μία ερώτηση προς έναν από τους εμπειρογνώμες, παρακαλώ, ο καθένας. <laughs> Θα προσπαθήσω, αλλά δεν τα καταφέρω. Γιατί έχω μια γενική ερώτηση. Δεν αγαπούν όλοι την παγκοσμιοποίηση και την παγκοσμιοποιημένη αγορά. Στο Ταβό έγινε μια πολύ αυστηρή δήλωση από τον Γάλλο Πρόεδρο και θα ήθελα να σας ρωτήσω όλους εσάς το εξής. Παγκοσμιοποίηση είναι απειλή στις ευρωπαϊκές με μια ψηφιακή ναι, είπε και εσείς ότι οι ευέλικτες ε, αγορές απασχόλησης το είπατε εδώ για το «Hard and fire το να προσλαμβάνει και να απολύει κανένα έτσι ελεύθερα, αυτό είναι μια αμερικανική πρακτική. Δεν είναι ευρωπαϊκή πρακτική αυτό. Βρισιά είναι σχεδόν. Λοιπόν, η ερώτηση προ τον κύριο Μπράουνερ, γιατί είσαστε και δύο Σουηδοί. Ε, αλλά και εσύ έχει μια ερώτηση. Παρακαλώ. Λέει η κυρία Σπίλμπορν. Στην Ουελία πάνω από το 90% των εργαζομένων είναι σε ΜΜΕ. Φαίνεται ότι ορισμένε από τι ε, ΜΜΕ έχουν ξεπεράσει την κρίση πιο καλά από τι μεγάλε εταιρείε που απολύσαν τόσο πολλού εργαζομένου. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν τεράστια προβλήματα για την δαδιολόγηση και οι καινούργιε επιχειρήσει είναι σχεδόν αδύνατο να βρουν το κεφάλαιο που χρειάζονται από τι τράπεζε. <clears throat> Από την άλλη μεριά έρχονται τράπεζε και ε, μου χτυπάνε την πόρτα και μου λένε μήπως μπορείτε να μας βοηθήσετε που έχει μειωθεί η ζήτηση κεφαλαίων. Ποιο θα πρέπει να είναι το χρηματοπιστωτικό μέσο που θα έχουμε κατά νου για να βοηθήσουμε τις ε, ΜΜΕ. Θα μπορούσατε να φανταστείτε παραδείγματος χάρη κάποια ταμεία για ε, κεφάλαια κινδύνου ή κάποιες δυνατότητες swap σε περιπτώσεις κρίσης. Τι. Ευχαριστώ, ρε Πρόεδρος. Κυρία Νοβάκ, θα απαντήσει αυτή την ερώτηση, αλλά ένα τρίτο συνάδελφο, Χάιντς. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Όλοι οι πολιτικοί βέβαια έτσι λένε. Θέλω να υποβάλω την ερώτησή μου στον κύριο Σράγιο. Έχουμε ένα παρόμοιο πρόβλημα. Έχουμε και εμείς πριν ένα παρόμοιο πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα των ΜΜΕ είναι ότι έχει σταματήσει η ροή του κεφαλαίου. Δεν πληρώνονται, αλλά από την άλλη μεριά έρχεται το κράτος και του ζητάει ε, φόρους ε, και διάφορες άλλες φορές. Ε, κάπου υπάρχει εδώ ένας ε, φαύλος κύκλος. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να υπάρξει κάποια ευρωπαϊκή ανεμενόπιση ή είναι ένα πρόβλημα συγκεκριμένη χώρα. Παρακαλώ. Κύριε Σπλαβέλ. Η παγκοσμιοποίηση ξέρετε ότι η παγκοσμιοποιηση ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Έχει σταματήσει κάπως, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα ξαναξεκινήσει. <clears throat> Κατά πόσο αυτό απειλεί τις ΜΜΕ, όχι θα έλεγα του αντίον, δημιουργεί πολλές ευκαιρίες για τις εταιρείε αυτές. Αλλά κατά πόσον αυτές οι ευκαιρίες θα μπορέσουν να μετατροπούν σε επιτυχείς ιδέες επιχειρησιακές, θα εξαρτηθεί πάρα πολύ από τις αποφάσεις των πολιτικών μας. Βάσει αυτών των τομέων πολιτικής που αναφέρα. Είναι σημαντικό να προχωρήσουν εδώ οι ΜΜΕ, αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε ανάπτυξη χωρίς απασχόληση. Okay. Novak. Well, as regards um, what kind of σε ό,τι αφορά τι είδους χρηματοδότηση θα πρέπει να διευκολύνεται. Μα χρηματοδότηση για κάθε είδους επιχείρηση. Ή χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ακόμα. Θα συμφωνούσα με τον κύριο Μπράουνερ Χέλμ ότι ε, το σημαντικότερο σε περιόδους κρίσεων είναι οι μετοχές και οι εγγύησεις. Και θα πρέπει να αναπτυχθεί αυτό, με ιδιωτικά κεφάλαια δηλαδή, ε, και εγγύησεις. <clears throat> E σε σχέση με την ερώτηση που θέσατε και που είναι κοινό το θέμα για τις χώρες μας, δεν μπορούμε να απαιτήσουμε από τις επιχειρήσεις αυτό που δεν έχουν. Και όσον αφορά την καθυστέρηση των πληρωμών, και ότι όποιος ε, ε, καθυστερεί, απαιτεί ε, τόκους για την καθυστέρηση των ε, πληρωμών. Ναι, να, πρέπει να τα πληρώνει, αλλά να τα πληρώνει και το κράτος άμα καθυστερεί να πληρώσει. Τώρα, μέσω της τράπεζας, άμα το κράτος δεν το κάνει όσον αφορά την, τον, τον, τον ΦΠΑ, ΦΠΑ, θα πρέπει οι επιχειρήσεις να μπορούν να πληρώνουν το ΦΠΑ με μικρές ε, ε, χαμηλούς τόκους που να είναι ανεκτοί για να μπορούν κατά κάποιο τρόπο άμεσα να, να λειτουργήσουν. και θα μπορούσε με τη σειρά του το κράτος ε, να χρεωθεί, να πληρώσει τις μικρές επιχειρήσεις. Το κράτος είναι υποχρεωμένο να πληρώσει τις τράπεζες με τη σειρά του και να μην υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις επικαθυστερήσεων ε, που εμποδίζουν όλους τους άλλους. Ναι. Υπάρχει μια σημαντική ερώτηση που έθιξε ο κύριος ε, Σμιτ, δηλαδή το hard and fire. Δεν νομίζω πως χρειάζεται να αντιγράψουμε το σύστημα των ΗΠΑ, αλλά είναι πολύ σημαντικό στοιχείο στο να διασφαλίσουμε ότι θα, υπάρχουμε, θα έχουμε μια οικονομία που είναι αναγκασμένη να μεταρρυθμιστεί. Η μεταρρύθμιση είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της ευημερία και για την ροή των πόρων σε περιοχές με μεγαλύτερη παραγωγικότητα και που δηλαδή μπορεί να βρίσκεται το μέλλον. Και πάλι τα, οι θεσμοί της αγοράς της εργασίας, η εκ νέου κατάρτιση, αυτό είναι το θέμα. Πρέπει δηλαδή να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο. Και δύο σοσιαλίστες τώρα τέλος, η κυρία Άλβαρες και η κυρία Σάρη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους εισηγητές μας για τις παρεμβάσεις τους. Ένα θέμα που όλοι γνωρίζουμε και θέτουμε είναι οι δυσκολίες στη χρηματοδότηση και στη δανειοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και θα ήθελα να ρωτήσω συγκεκριμένα την κυρία Νόβακ σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Χρειάζεται καμιά αλλαγή στην αρμοδιότητά της, στις εξουσίες της, στη λειτουργία της για να αποδίδει καλύτερα και να χρηματοδοτεί, να δανειοδοτεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ κυρία Γιακονσάρη. Στη Φιλανδία Εάν μια εταιρεία έχει μια πολύ καινοτόμα ιδέα και πολύ ενδιαφέρουσα, χρηματοδότηση θα βρει. Γιατί είπαν όλα τα κρατημέλη ότι θέλουν να προωθούν την καινοτομία και την εφευρετικότητα. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Όταν κάποιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα πρόσβασης, δεν έχουν αυτή τη γέφυρα, θέλετε, ε, και δεν έχουν τη δυνατότητα να βγουν από την κρίση και να γνωρίσουν καλύτερες μέρες. Αντιμετωπίζουν ένα μεγάλο πρόβλημα και θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο σε σχέση με αυτά που ρώτησαν συνάδελφοι. Κάπως διαφορετικά. Πώς θα μπούμε σε αυτή τη νέα στρατηγική που λέμε του 2020 του 2020, 2020 πώς θα διευκολύνουμε ε, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. σε ποιο, ποια ρωτάτε, όποιον μπορεί να την απαντήσει καλύτερα, λέει η κυρία Γιακονσάρη. Η κυρία Νόβακ. Εγώ δεν είμαι σε θέση να αξιολογήσω ολόκληρη την πολιτική ε, δανειοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Απλώς θέλω να πω ότι σε περιόδους κρίσης είναι σημαντικό να αναπτύσσει κανείς όλες αυτές τις μορφές χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και προς τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Και βεβαίω απομένει ακόμα πολλή δουλειά. Κύριε Μπρόν, θέλουμε να προσπαθήσετε κι εσείς να απαντήσετε στην τελευταία ερώτηση. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Σημαντικό αυτό που λέτε και στη Σουηδία βλέπουμε ότι το 1 τρίτο περίπου των μικρών επιχειρήσεων ε, κάνουν περικοπές στην έρευνα και στην ανάπτυξη, δηλαδή κυρίως στην ανάπτυξη στο εσωτερικό των εταιριών. Μα κανονικά από εκεί θα πρέπει να προέλθει η μελλοντική τους ανταγωνιστικότητα και είναι πρόβλημα. Οι μικρές επιχειρήσεις ε, που ήδη εστιάζονται στην έρευνα και την ανάπτυξη αμυγός, γιατί αυτό είναι ο δρόμος προς τη μελλοντική τους επιτυχία, θέλουν να συνεχίσουν σε αυτό το δρόμο. Και αυτοί είναι εκείνοι που βρίσκουν ε, τις ε, λαμπρές ιδέες, φαίνες ιδέες που είπατε κι εσείς. Πώς το χειρίζεσαι αυτό από πλευράς πολιτικής είναι πολύ δύσκολο. Γιατί πώς θα ξεχωρίσουμε τις καλές από τις κακές ιδέες ανάλογα με τον επενδυτή αξιολογείται κάθε ιδέα με διαφορετικό τρόπο και χρειάζεται ποικιλία επενδυτών, μια παλέτα ολόκληρη για να υποστηρίζουν αυτές οι επιχειρήσεις, όχι μόνο οι κυβερνήσεις. Εκεί θα πρέπει εμείς να γίνουμε καλύτεροι στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους τρεις εξ ονόματος της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ που ήρθατε να μας μιλήσετε και να απαντήσετε ειλικρινά και στις ερωτήσεις μας. Ακολουθεί δεύτερο πάνελ και αλλαγή σκητάλης. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε με το δεύτερο πάνελ. που αναφερόμαστε στην ε, εξέλιξη πολιτικών αποφάσεων για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που παρουσιάστηκε στο προηγούμενο πάνελ. Χαίρομαι να σας παρουσιάσω δύο συμμετέχοντες. Έχετε τις λεπτομερείς, ε, λεπτομεριά βιογραφικά σημείωματα. Χαίρομαι που έχουμε και στο δεύτερο πάνελ μια κυρία, Ράνι Χελτεφόγγελε. Είναι σημαντικό γιατί πολλές φορές με κατηγόρησαν ότι δεν μπορούσαμε να έχουμε μια γυναίκα εδώ απάνω στο βήμα. Δύο είχαμε σήμερα λοιπόν. Ράνι Χελτεφόγγελε είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Λέβεν. Μετά έχουμε τον Γιάννη Φίμερ στην Ευρωπαϊκή Ένωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και υπεύθυνο για την οικονομική και εφαρμογική πολιτική και τρίτον έχουμε εδώ τον Γιώργο Ιωαννίδη που είναι Visiting Fellow στο Τμήμα Πολιτικών και Διεθνών Μελετών στο Cambridge. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ. Θα σας ακούσουμε πολύ ενδιαφέρον. Κυρία Καθηγήτρια, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Θα ήθελα να σας μιλήσω για το εξής. Τα εξής τέσσερα θέματα. Ε, εξασφάλιση της σημασίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την περίοδο μετά την κρίση και μια συγκεκριμένη κατηγορία που είναι ιδιαίτερα καινοτόμη. Στη συνέχεια θέλω να αποδείξω ποιο είναι ο αντίκτυπο της κρίσης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και είναι ευκαιρία γι' αυτό. Το τρίτο, ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε διαρθρωτικές αδυναμίες των μικρομεσαίων να αναλάβουν αυτό το ρόλο και το σημαντικότερο αν υπάρχει ε, ρόλος για κυβερνητικές παρεμβάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αυξηθεί ε, και να τονωθεί ο ρόλος των μικρομεσαίων. Λοιπόν, γιατί είναι τόσο σημαντικές για την ανάπτυξη οι μικρομεσαίες. Αν αναλύσουμε το συναλλικό ε, και τη συναλλική ανάπτυξη που είναι οι πιο ε, παραγωγικές εταιρείες, η έξοδος των λιγότερων παραγωγικών και των σημειογόνων, ε, ε, αυτή λοιπόν τη διαδικασία εισόδου-εξόδου από την αγορά ε, είναι πολύ σημαντικό να το αναλύσουμε για να δούμε ποια είναι η διαφορά μεταξύ μιας επιτυχούς και μιας αποτυχημένης οικονομίας στην Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο. Και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι στην καρδιά ακριβώς αυτού του στοιχείου γιατί μπαίνουν με μεγάλους ρυθμούς, βγαίνουν με μεγάλους ρυθμούς και αναπτύσσονται με μεγάλους ρυθμούς. Ε, κάνουν ε, πειράματα με νέες ε, προσεγγίσεις με καινοτομία στην Ευρώπη. Λοιπόν, σε αυτή τη διαδικασία της εναλλαγής οι νέες εταιρείες, οι καινοτόμες είναι πολύ σημαντικές και είναι μικρομεσαίες. Αν υπάρχουν σημαντικά εμπόδια και φραγμοί για να βγαίνουν από την αγορά αυτέ οι επιχειρήσει, αυτό είναι αρνητικό, γιατί εμποδίζει αυτή την κυκλοφορία, την, έσοδο, την είσοδο και την έξοδο και την ανάπτυξή του και τη δυναμική του. Ε, είναι οι άμεσε επιπτώσει, αλλά και έμεσα μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο οι μικρομεσαίε, διότι ε, τονώνουν την πιο καινοτόμο προσέγγιση και συμπεριφορά και των μεγαλύτερων εταιριών με τη δική του παρουσία μικρομεσαίε και μπαίνοντας στην αγορά λοιπόν ε, δημιουργούν ε, κίνητρα για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και αυτές περισσότερο. Έχουμε λοιπόν και άμεση και έμεση συμμετοχή των μικρομεσαίων. Και όλα αυτά επηρεάζουν σοβαρά την περίοδο μετά την κρίση. Τι θα μπορούσε λοιπόν να επαρεμποδίσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αυτό ε, δείχνει τη σημασία της ε, πρόσβασης στη ότι είναι ειδικό φραγμός και ειδικό εμπόδιο για τις ε, νέες επιχειρήσεις με νέα στελέχη, με καινοτόμα και αυτοί οι νέοι επιχειρηματίες έχουν τη μεγαλύτερη δυσκολία πρόσβασης σε κεφάλαιο. Το επόμενο που θέλω να πω είναι ότι η σημερινή κρίση ε, είναι επιζήμια πολύ και ε, για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γνωρίζουμε από τις έρευνες ότι επιχειρηματίες που καινοτομούν και είναι ηγετικές επιχειρήσεις και είναι και μπροστά από την εποχή τους, δύο χρόνια περίπου. Λοιπόν, αυτό το επιχειρηματικό πνεύμα είναι εκείνο που δίνει μια θετική όθηση στην οικονομία και πυροδοτεί και την ανάκαμψή της. Οι εταιρείε λοιπόν που έχουν μεγαλύτερες δυσκολίες πρόσβασης γιατί είναι υψηλού κινδύνου πλήττονται ιδιαίτερα από μια χρηματοπιστωτική κρίση. Ιδιαίτερα σε περιοχή ύφεση με μεγάλα ποσοστά πτωχεύσεων. Και αυτές οι νέες εταιρείες, οι καινοτόμες, έχουν ένα προφίλ υψηλού κινδύνου, με μεγάλο κίνδυνο πτώχευσης και σε μεγάλο βαθμό ε, εξαρτώνται από εξωτερική χρηματοδότηση. Και είναι διπλό το πρόβλημα, γιατί έχουν μεν μεγάλη ανάγκη χρηματοδότηση, αλλά ταυτόχρονα και μεγάλο κίνδυνο να πτωχεύσουν. Ε, τώρα, σε ποιο βαθμό υπάρχει ειδικό πρόβλημα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ένωση και πώς εμποδίζει να παίξουν το ρόλο του στον αναπτυξιακό. Τι συνέβαινε πριν από την κρίση, ανεξάρτητα με την κρίση. Το πρόβλημα με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ότι δεν έχουμε αρκετές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ακούσαμε ήδη αρκετά που στοιχειοθετούν ότι είναι αρκετές επιχειρήσεις στον αριθμό, αλλά ποιο ρόλο μπορούν να παίξουν και αναπτυξιακό ρόλο εννοώ. Μα δείχνουν λοιπόν τα στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειε, αλλά στην Ένωση έχουμε μικρότερη κυκλοφορία εισόδου-εξόδου από την αγορά εταιριών καινοτόμων στις νέες τεχνολογίες και τέτοιους κλάδους. Και αυτό συνδέεται με το γεγονός ότι μας λείπουν αυτά τα ε, ε, ταλέντα, αυτοί οι νέοι επιχειρηματίες, οι πιο καινοτόμοι και οι πιο ε, εφευρετική. Λοιπόν, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε αυτή την είσοδο και έξοδο εταιριών και στις ε, εταιρείε που είναι ιδιαίτερα ψηλής καινοτομία και ανάπτυξη. Για ποιο λόγο δεν έχουμε αυτή την καινοτομία και αυτές τις εταιρείε στην Ευρώπη. γιατί οι αγορές μας δεν είναι ε, ολοκληρωμένες όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ε, έχουμε και εμπόδια ε, όχι μόνο στην είσοδο αλλά και στην έξοδο ζημιογόνων εταιριών από την αγορά και έτσι δεν δημιουργείται ε, χώρος για να μπουν οι, κοινο, καινοτόμες και οι ε, πιο σύγχρονες. Γενικά το σύστημα στην Ευρώπη ε, δεν ευνοεί την καινοτομία και οι μικρομεσαίες συμβιούν με μεγαλύτερες εταιρείες ε, και εμφανίζεται μεγαλύτερη βραδύτητα στην ανανέωση, στην καινοτομία ε, και δεν αλλάζει το σύστημα, δεν ανανεώνεται. Είναι πιο κατακαιρματισμένες οι αγορές ως προς το κίνδυνο και τα προϊόντα και δεν δίνονται μεγάλα κίνητρα για την καινοτομία. και υπάρχουν ε, προβλήματα στην πρόσβαση, στα κεφάλαια, στη δανειοδότηση. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό. Για τις νέες εταιρείες και τους νέους επιχειρηματίες είναι πρόβλημα και αυτό ήταν πρόβλημα και από το παρελθόν και εντάθηκε και οξύνθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης. Τώρα, ε, πώς ε, μπορούν να δράσουν οι κυβερνήσεις, τι ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν. Οι οικονομικές αναλύσεις ε, δείχνουν ότι δεν ξέρουμε στην Ευρώπη τι αποδίδει και τι δεν αποδίδει. Θα μπορούσαμε να πούμε τι δεν πρέπει να κάνουμε περισσότερο παρά ε, το τι να κάνουμε. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και μεγάλος πειρασμός σε περιόδους κρίσεων δεν θα πρέπει να αφήσουμε προβληματικές εταιρείες σε προβληματικούς τομείς να ε, λειτουργούν. Γιατί έτσι ε, παρεμποδίζεται η είσοδος κάποιων άλλων καινοτόμων εταιρείων στην αγορά. Ε, δεν χρειάζεται τέτοια προστασία. Θα πρέπει να υπάρχουν ειδικά κατόφλια στις ε, ε, νομοθεσίες lock-in για τις μικρομεσαίες και θα πρέπει να αποφεύγουμε τις λύσεις ad hoc γιατί ε, δεν βοηθούν. Αυτά είναι τα αρνητικά βεβαίως, τα, τα θετικά. Αυτό που προτείνουμε να κάνουμε ενδεχομένω είναι ε, η αποκατάσταση των χρηματαγορών γιατί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι πολύ σημαντικό. Τι σημαίνει αυτό. Να είμαστε βέβαιοι ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέα θα δίνει δάνεια με όρους ανταγωνιστικούς ε, και με αηφόρο ανάληψη του κινδύνου. Βεβαίως, πρόβλημα υπήρχε, είπαμε και πριν από την κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις μικρομεσαίες, γι' αυτό η πολιτική αυτή είναι λίγο πιο μακροχρόνια. Και αυτό έχει να κάνει με τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για την καινοτομία και την ανάπτυξη από τις ίδιες μικρομεσαίες. Τι σημαίνει αυτό. Να λειτουργεί η αγορά με τρόπο πιο αποτελεσματικό πιο ολοκληρωμένο, να αλλάξει το πτωχευτικό δίκαιο. Η ολοκλήρωση των χρηματαγορών, ιδιαίτερα της αγοράς κεφαλαίων κινδύνου, βελτίωση στο φαρολογικό σύστημα και μείωση ε, των διοικητικών ε, εμποδίων και φραγμών. Αυτά είναι ίσως γενικότερα ε, και περιγράφουν γενικές πολιτικές και δεν αφορούν συγκεκριμένα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα, χρειάζεται ε, ειδική παρέμβαση για τις μικρομεσαίες, ναι. Χρειάζεται ειδική πολιτική που να προωθεί την καινοτομία και να αντιμετωπίζει τα ιδιαίτερα προβλήματά τους. Και υπάρχουν και υποκατηγορίες μικρομεσαίων και εντός των κατηγοριών αυτών διαφορετικά τα προβλήματα και διαφορετική φραγμή και τα εμπόδια και γι' αυτό χρειάζονται ειδικά εργαλεία μικροπιστώσεις για τις πολύ μικρές εταιρείες. για να έχουν πρόσβαση πολύ μικρές καινούριες καινοτόμες ε, εταιρείε. Ε, χρειάζεται μια πολιτική σχεδιασμένη ειδικά για τις μεσές. Και επειδή τελειώνει ο χρόνος μου, πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε ειδικά μέσα για νέα στελέχει νέες και καινοτόμε για να μπουν στην αγορά. Για τη συγκεκριμένη λοιπόν υποκατηγορία το σημαντικότερο και πρώτο είναι Θα πρέπει να υπάρχει ένα οικοσύστημα ήδη στην οικονομία καινοτομία που να λειτουργεί σωστά. Για να μπει ένα οποιοδήποτε καινούριο στοιχείο πρέπει να βρει πρόσφορο έδαφο. Πέρα από αυτό όμως χρειάζονται και ειδικά μέσα για να αντιμετωπίζουν ειδικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι νέες καινοτόμες επιχειρήσεις. Προηγουμένως είπα ότι η πρόσβαση στις πιστώσεις και οι περιορισμοί είναι πάρα πολύ κρίσιμη για τις εταιρείες αυτές. Λοιπόν, ειδικά εργαλεία που να αντιμετωπίζουν ε, τα οικονομικά προβλήματα αυτών των συγκεκριμένων εταιρεών, ειδικά προγράμματα επιδοτήσεων, που να ανταμείβουν ε, την ανάληψη κινδύνου σε ε, αυτές τις καινοτόμες εταιρείε. Έχουμε κάνει και ειδική μελέτη και ειδική πρόταση. Και για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι επίσης πολύ δύσκολο να έχουν καλή προστασία των πνευματικών τους δικαιωμάτων όταν καινοτομούν και κάνουν ε, παρεμβάσεις με νέες εφηβρέ. Σας είπα ότι αυτές είναι ε, κάποιες λεπτομέρειες, αλλά επειδή δεν έχω χρόνο την αφήνω τη διαφάνεια στην άκρη και έρχομαι στην τελευταία. Οι περισσότερες πολιτικές ανάπτυξη των μικρομεσαίων που συζητούμε είναι περισσότερο σε επίπεδο κρατών μελών. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βέξει το ρόλο της εκεί, με την ενιαία αγορά βεβαίως που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ε, και οι χρηματαγορές ε, βεβαίω προχωρούν σε ενιαία αγορά, οι κρατικές ενισχύσεις και ο ανταγωνισμός και πώς μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε τις διαφόρες μικρομεσαίες και επίσης η Ένωση μπορεί να παίξει ρόλο ελέγχοντας τις αγορές και τις πολιτικές για να έχουμε τις βέλτιστες πρακτικές και να διδάσκεται ο ένας από τον άλλον. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Και που ε, σας απασχολούν τα προβλήματα των ΜΜΕ δηλαδή διάρκεια της κρίσης. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να μιλήσω αγγλικά, γιατί έτσι έχω προετοιμάσει τις ε, διαφάμες. να αναφέρθηκαν σε πάρα πολύ καινοτόμε εταιρείε που είναι πάρα πολύ σημαντικέ, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε όταν συζητάμε την πολιτική για τη ΜΜΕ, το 99, κάτι των επιχειρήσεων δεν είναι ιδιαίτερα καινοτόμε, Αλλά είναι παρόλα αυτά πάρα πολύ σημαντικέ, όχι μόνο για τη δημιουργία θέση απασχόληση, αλλά και όσον αφορά την κανονική καινοτομία. Είναι σαφές για όλους νομίζω ότι υπέφεραν από την κρίση η ΜΜΕ. και στον τομέα των οικοδομών στην αρχή και μεταξύ σε όλους τους οικονομικούς τομείς. Και θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις, η αύξηση δηλαδή της ανεργίας είχε επιπτώσεις στην ιδιωτική κατανάλωση και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι ΜΜΕ το 2010. Αυτό που θέλω να κάνω σήμερα είναι να σας δώσω μια πολύ σύντομη εικόνα διαφόρων τομέων πολιτικής που σχετίζονται άμεσα με τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Είναι σαφές, όπως το είπε συνάδελφος, τα περισσότερα από τα άμεσα μέτρα που λαμβάνονται από τις ΜΜΕ σχετίζονται με εθνικές περιφερειακές κυβερνήσεις. Υπάρχουν όμως και άλλα στοιχεία τα οποία βρίσκονται στο ευρωπαϊκό επίπεδο και όπου οι επιφάσεις που λαμβάνουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγγνώμη, ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν σημαντικές επιπτώσεις της ΜΜΕ. Το πρώτο που θέλω να φέρω είναι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, το δεύτερο είναι τα γενικά ε, προγράμματα ανάρρωσης και τέλος το θέμα του δημοσίου τομέα. Όσον αφορά το θέμα των μέτρων χρηματοδότησης, υπάρχουν προβλήματα. Στην αρχή, ε, οι τράπεζες είχαν προβλήματα για την χρηματοδότηση των δανείων στις ΜΜΕ λόγω προβλημάτων ρευστότητας. Αυτή η περίοδος έχει τελειώσει. Τώρα το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει αρκετό κεφάλαιο για να διευρυθούν οι γραμμές αυτές δυνατότητες. Και έχουμε λίγο πολύ το ίδιο πρόβλημα που είχαμε στη δεκαετία του 90, αλλά κυρίω το πρόβλημα για τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ είναι ότι εάν ξαναξεκινήσει να ανακάμπτεται η οικονομία, τότε θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί η ανάπτυξη αυτή. Γιατί αυτή τη στιγμή οι τράπεζες όσο πάει και περισσότερο δεν θέλουν ή δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν ε, διακυβευόμενα προγράμματα. Δεν είναι πια τα δάνεια αυτά το κατάλληλο χρηματοδοτικό ε, μέσο αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να μελετήσουμε τι θα πρέπει να κάνουμε για να αναπτυχθούν χρηματοπιστωτικά μέσα για τις ΜΜΕ που να επιτρέψουν να καλυφθούν κεφάλαια κινδύνου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Από πολλές αναλύσεις αγοράς ξέρουμε ότι τα ιδιωτικά κονδύλια κατά οποιονδήποτε τρόπο δεν ε, ε, λειτουργούν πάνω από τα 2 εκατομμύρια ευρώ χωρίς την δημόσια υποστήριξη. Και εδώ χρειάζεται μία λύση. Αυτό είναι μία πραγματική πρόκληση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των ΜΜΕ. Θα πρέπει να υπάρχουν οι σωστοί διαγωνισμοί. Και χρειάζεται καλύτερη σταθεροποίηση της αγοράς και αυτό δεν πρέπει να γίνει η βάρος της χρηματοδότησης των ΜΜΕ. Αν χρειαζόμαστε περισσότερα κεφάλαια, ίσως σε κάποιους άλλους τομείς. Θα πρέπει να υπάρχουν καλά συστήματα τραπεζών και βλέπουμε ότι οι χώρες που το έχουν αυτό είναι εκείνες που αντιμετωπίζουν την κρίση καλύτερα. και όχι εκείνες όπου οι ΜΜΕ εξαρτώνται για τη χρηματοδότηση του από μεγάλε εμπορικέ τράπεζε. Και η διακανόνιση της αγορά δεν θα πρέπει να ε, διακυβεύσει το σύστημα που λειτουργεί. Δεν θα επαναλάβω αυτά που ελέγχθησαν από τους συναδέλφους πριν από μένα. Αλλά το επόμενο στοιχείο στο οποίο θέλω να αναφερθώ είναι γενικά τα προγράμματα ανάκαμψης. Και βλέπουμε ότι υπάρχει όσο πάει και περισσότερο ζασμός για τις λεγόμενες ε, στρατηγικές εξόδου, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το πώς θα γίνει εξόδος από τα συστήματα ανάκαμψη. Θα πρέπει οι επιχειρήσεις να ξέρουν πώς θα λειτουργήσει αυτό σε ένα-δύο χρόνια για να είναι έτοιμες. Είναι απαράδεκτο για τις ΜΜΕ να μην ξέρουν τι θα γίνει γιατί βλέπουν ότι μεγάλες εταιρείε εξακολουθούν να χρηματοδοτούνται από το κράτος για να προστατεύσουν πεπαλαιωμένες δομές. Και ξέρουμε από ότι όσο πιο περισσότερο χρόνο χρηματοδοτείται σε μια κρίση μια πεπαλαιωμένη δομή, τόσο πιο μεγάλο είναι το πρόβλημα στο μέλλον. Θα πρέπει τα χρήματα να χρησιμοποιηθούν για, τον, για το μέλλον για τη χρηματοδότηση ιδιωτικών επιδίσεων ιδιωτικής κατανάλωσης και όχι μέσω της δημόσιας ε, κατανάλωσης. Τελευταίο σημείο. Δημόσιος τομέας. Θα ξεκινήσουμε με την ε, στρατηγική 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020. Στην αρχή όταν το εξτάσαμε μας έκανε φοβερή εντύπωση ότι Όλο αυτό το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2020 δεν αναφέρεται καθόλου στο θέμα της ποιότητας και της ικανότητας των ε, διακανονιστών και είναι σαφές για όλους μας ότι η οικονομία αγοράς χρειάζεται βέβαια καλό διακανονιστικό πλαίσιο και αν υπάρχουν αυτοί οι διακανονιστές που είναι ανεξάρτητοι και αρκετά ισχυροί για να ε, περιβάλλουν τον οργανισμό θα υπάρχει ένα πρόβλημα παντού στον τομέα των μεταφορών και σε άλλου. Αυτή είναι μια πτυχή. Μια άλλη πτυχή είναι οι δημόσιε υπηρεσίε. Οι φορολογούμενοι στο μέλλον και οι ΜΜΕ είναι ε, οι φορολογούμενοι και οι εργαζόμενοι όσους είναι οι περισσότεροι φορολογούμενοι της Ευρώπης. Δεν θα μπορέσουν να δεχθούν να πληρώνουν τους φόρους εάν βλέπουν τα χρήματα αυτά δεν δαπανούνται αποτελεσματικά. Δεν είναι αρκετά τα κλπ. κλπ. Υπάρχουν χώρες που υπάρχουν υψηλά επίπεδα φορολόγησης και άλλες η αποδοχή είναι ανώτερη γιατί ε, η αποτελεσματικότητα του δημοσίου τομέα είναι καλύτερα από τις άλλες. Δεν θα αναφέρω τώρα συγκεκριμένε χώρες, αλλά ονονοητό. το θέμα της εξόδου από την κρίση θα πρέπει να τονίζει ακόμα περισσότερο το δημόσιο προπολογισμό. Ε, οι πολίτες δεν θα δεχθούν τις επιστροφές αυτές παρά μόνο εάν έχουν την εντύπωση ότι τα χρήματα χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά. Μετά πρέπει να σκεφτούμε το, την αρχή του Think Small First το SBA έχει δίκιο ο κύριο ότι πολλά από αυτά θα πρέπει να γίνουν σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπορούν να γίνουν πολύ περισσότερο για να α, παρουσιαστούν οι κύριε αρχέ όσον αφορά την αξιολόγηση των επιπτώσεων, στο αφορά διαβούβορση. Πράγματα που τα έχουν ζητήσει οι ευρωπαϊκέ αρχέ ήδη. Δεν θέλω να επισέλθω στι λεπτομέρειε εδώ, αλλά τα θεσμικά όργανα τη Ευρώπη θα πρέπει να αποδείξουν ότι ακολουθούν και σέβονται αυτέ τι αρχέ. Αυτά με δύο λόγια μόνο, μια σύντομη παρουσίαση, λόγω του περιορισμένου του χρόνου που είχαμε. Αν θέλετε να διαβάσετε κάτι παραπάνω για τους τομείς αυτής, θα δείτε στα slides αυτά ε, ένα link που να παρουσιάζει ακριβώς ένα 20 σελίδο κείμενο για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επόμενα πέντε χρόνια και μπορούμε να σας δώσουμε και λεπτομέρειες θέλετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Χιμά. Ο κύριος Ιωαννίδης έχει το λόγο. Ε, φανταστείτε να έπρεπε να διαμορφώσετε μια πολιτική όσον αφορά την απασχόληση και να μην μπορούσατε μετά από τρία χρόνια να πείτε πόσες νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν. Αυτή όμως είναι περίπου η κατάσταση που ισχύει με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ίσως ένα από τα πιο μόνιμα χαρακτηριστικά και σημαντικά προβλήματα για όσους διαμορφώνουν πολιτική είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία. Η κατάσταση δεν είναι ίδια για όλες τις χώρες. Κάποιες βρίσκε, σε κάποιες χώρες υπάρχει ε, αρκετό στατιστικό υλικό, σε κάποιες άλλες δεν υπάρχει καθόλου. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι ένα από τα ζητήματα, τα τεχνικά πλήν όμως πάρα πολύ σημαντικά που θα πρέπει να γίνει, είναι να μπορέσει να φτιαχτεί επιτέλους μια μόνιμη και σταθερή βάση στατιστικών δεδομένων σε σχέση με την επιχείρημα... Ναι. Σε σχέση με την επιχειρηματική δημογραφία. Τώρα, ένα από τα προβλήματα που ήθελα να θίξω είναι το πρόβλημα της κοινωνικής προστασίας του μικρού επιχειρηματία. Ενώ τα περισσότερα κράτη έχουν αναπτύξει κάποιο, συστημα, κάποιο τύπου συστήματα κοινωνικής υποστήριξης για κάποιον εργαζόμενο, για παράδειγμα, που χάνει τη δουλειά του, αυτή δεν είναι πάντα η περίπτωση όσον αφορά τους μικρούς επιχειρηματίες μια οικογενειακής επιχείρησης η οποία κλείνει. Δεν θέλω να συγκρίνω προφανώ τον πόνο των ανθρώπων που βρίσκονται άνεργοι, είτε ήταν πριν εργαζόμενοι, είτε ήταν πριν επιχειρηματίε. Αυτό όμω που θέλω να πω είναι ότι η έννοια, αν θέλετε, τη δημιουργική καταστροφή που οι οικονομολόγοι μα αρέσει πάρα πολύ, είναι μια χρήσιμη έννοια για να μπορέσει η οικονομία να προσαρμοστεί στις νέε συνθήκε, προποθέτει όμω ένα ισχυρό σύστημα κοινωνική προστασία, το οποίο να μπορεί να διαχειριστεί το κόστο τη αλλαγή στο νέο μοντέλο και ειδικά όσον αφορά τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τις οικογενειακές επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους, συχνά αυτά τα συστήματα είναι υποανεπτυγμένα. Σε αυτό το πεδίο νομίζω ότι οι οργανώσεις των μικρών επιχειρήσεων και τα επιμελητήρια θα μπορούσαν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο, στο μέτρο βέβαια που είναι αρκετά δυνατά και με οικονομικούς και με οργανωτικούς όρους, συχνά όμως θα πρέπει να μπορέσουν να υποστηριχθούν και από το κράτος με ένα προβοκατόρικο, αν θέλετε, τρόπο, θα έλεγα ότι μέσα σε μια περίοδο κρίσης και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως όλοι οι υπόλοιποι, θα πρέπει να σκεφτούν όχι μόνο και αποκλειστικά με όρους ανταγωνιστικότητας, αλλά και με όρους αλληλεγγύης. Τώρα, όταν το 99, σε μια οικονομία που το 99% των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι προφανές ότι η οικονομική κρίση σημαίνει και κρίση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό μου δίνει τη δυνατότητα να κάνω ένα σχόλιο μακροοικονομικού, αν θέλετε, χαρακτήρα όσον αφορά τις, ε, το επόμενο διάστημα. Είναι γεγονό ότι το πιο άμεσο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πολύ μικρέ επιχειρήσει είναι το ζήτημα τη πρόσβαση στη χρηματοδότηση εν μέσω τη ε, οικονομική κρίση. Δεν είναι όμω το μόνο. Όπω ακόμα και ο, όπως ο ΣΑ ανέδειξε σε πρόσφατη μελέτη όσον αφορά την, με θέμα την κρίση και τι μικρομεσαίες επιχειρήσει, οι πολύ μικρέ επιχειρήσει αντιμετώπισαν ένα διπλό σοκ. Το πρώτο αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και το δεύτερο αφορά μια δραστική μείωση της ζήτησης για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Το ενδιαφέρον στοιχείο εδώ πέρα που θέλω να τονίσω είναι ότι αυτή η μείωση της ζήτησης ήταν το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πριν την κρίση. Το Μάιο του 2007, στο Ευρωβαρόμετρο με θέμα μικρομεσαίες επιχειρήσεις και με δείγμα 17.000 μικρές επιχειρήσεις από όλη την Ευρώπη, η πρόσβαση, το πρόβλημα της πρόσβασης στη χρηματοδότηση ήταν μόλις το έκτο πιο σημαντικό ζήτημα, το οποίο και αφορούσε το 21% των επιχειρήσεων. Το πιο σημαντικό πρόβλημα, το οποίο δήλωσε το 46% των μικρών επιχειρήσεων, ήταν η μειωμένη αγοραστική δύναμη των πελατών τους. Ακόμα πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι άμα πάμε στις μεγάλες επιχειρήσεις, δηλαδή αυτές που απασχολούν πάνω από 250, 250 ε, υπαλλήλους, το πρόβλημα της μειωμένης αγοραστικής δύναμης αφορούσε μόνο το 29% των επιχειρήσεων. Εδώ δηλαδή το μέγεθος μετράει. Όσο πιο μικρή είναι μια επιχείρηση, τόσο πιο προσανατολισμένη είναι στην εσωτερική αγορά, τόσο πιο περιορισμένες είναι οι αγορές στις οποίες μπορεί να πουλήσει τα προϊόντα της. Αυτό που θέλω να πω για να καταλήξω είναι ότι υπάρχει ότι έχει έρθει ίσως η στιγμή να ξαναδούμε τα βασικά χαρακτηριστικά τα οποία ε, διαπερνούν την οικονομική, μας, ε, την οικονομική πολιτική. Είναι ένα στοιχείο το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με συνέπεια έχει τονίσει τα τελευταία χρόνια ότι πρέπει να αποκατασταθεί η ενότητα της δημοσιονομικής και της νομισματικής πολιτικής. Δεν μπορούμε να έχουμε μια νομισματική πολιτική που να στοχεύει αποκλειστικά και μόνο στην ε, μείωση του πληθωρισμού εκτός των άλλων με δεδομένο ότι ο βαθμός χρησιμοποίησης του βιομηχανικού δυναμικού είναι μόλις το 70% και η ανεργία είναι στο 10% σημαίνει ότι ο κίνδυνος για τον πληθωρισμό είναι μάλλον υπερεκτιμημένος και στηρίζεται και οι επιστημονικές του βάσεις επερωτούνται έντονα. Ωστόσο, η πολιτική, και με αυτό κλείνω, η πολιτική την οποία προτείνω ε, προϋποθέτει και, και κάποια εργαλεία. Νομίζω τα άμεσα μέτρα θα ήταν ε, αν τι άλλο, η, έκδοση, η, η, σκέψη γύρω από την έκδοση ενός ευρωπαϊκού ομολόγου, προκειμένου να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί μια τέτοια πολιτική στήριξη και των μικρών, μεσών επιχειρήσεων και προφανώς η ανάπτυξη της, ε, του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Η αύξηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές μας και ερχόμαστε στις ερωτήσεις. Αρχίζουν και πάλι από τους συντηρητικούς. Μπένσον και Ότμαρ Κάρας. Ότμαρ, άρχισε εσύ και μετά βλέπουμε. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω το εξής. Θα χαιρόμουν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να το χαρακτηρίζατε ως χριστιανοδημοκράτες και όχι πάντα συντηρητικού στη γωνία. Εν πάση περιπτώσει, δεν, είκουμε όλοι στην ίδια αυτή κατηγορία. Έρχομαι τώρα σε ερώτηση μου. Ερώτηση πρώτη. Ποιο δυναμικό ε, έγκυται στην ελευθερία παροχής ε, υπηρεσιών για τις υπηρεσίες και τις επιχειρήσεις που τις παρέχουν. Η οδηγία για τις ε, υπηρεσίες είναι καλή, επαρκή, πού υπάρχει ακόμα εμπλοκή και εφαρμόζεται σωστά. Και δεύτερη ερώτηση, όλοι μιλάμε για καινοτομία. Εσείς πώς το μετράτε. κύριε Χιούμερ, ή και οι επιστήμονες. Πώς τη μετράτε την καινοτομία, δηλαδή για να αξιολογήσουμε την καινοτομία, θέλουμε ένα ράστερ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το τρίτο σημείο, θέλω και ένα benchmark, ένα σημείο αξιολόγησης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι ανταποκρίνεται στα δικά σας ιδεώδη για τη χρηματοδότηση, για την επένδυση και για τη διοικητική απλούστευση και την αύξηση της απασχόλησης. Πού είναι ο κατάλογος των συγκρίσεων και της συγκριτικής αξιολόγησης του benchmarking για να μπορέσουμε να προσανατολιστούμε. Θυμάστε όταν συζητούσαμε το πακέτο για τις τράπεζες ε, ε, και την ανταγωνιστικότητα. Ε, μήπως χρειαζόμαστε και ένα πακέτο για τις μικρομεσαίες, για την ανάληψη της αστικής ευθύνης, για το διαχωρισμό των κρατικών ενισχύσεων με τις μελλοντικέ επενδύσεις και τις επενδύσεις που είναι στραμμένες στο μέλλον. Εγώ έχω υποβάλει λοιπόν και τις τρεις ερωτήσεις και στους τρεις σας. Όποιος μπορεί να απαντήσει ε, καλύτερα, ας μου απαντήσει. Η πρώτη ερώτηση είναι προς τον κύριο Χιούμερ για την πράξη, η δεύτερη για την καινοτομία προς την καθηγήτρια την κυρία Φόγκλας και η τρίτη ερώτηση ίσως προς το νεότερο φίλο μας από το Κέμπριτζ, τον κύριο Ιωνίδη και ε, η επόμενη ερώτηση αποφασίστε ποιος θα την απαντήσει. Ο κύριος Χιούμερ, η οδηγία για την παροχή υπηρεσιών κανονικά θα πρέπει τέλη του έτους να έχει εφαρμοστεί και να έχει μεταφερθεί. Ξέρω ότι όλα τα κράτη-μέλη δεν εφαρμόζουν όπως θα πρέπει την οδηγία, αλλά είναι δύσκολο να πούμε από τώρα τι λειτουργεί καλά και τι δεν λειτουργεί. Η πρακτική εμπειρία με όλα αυτά τα συστήματα ε, υποστήριξης δεν είναι αρκετή για να την αξιολογήσουμε. Ακούσατε και προηγουμένως από την συζήτηση τι γίνεται στην Πορτογαλία και στη Γαλλία. Δηλαδή, από εθνικής απόψεως η ελευθερία υπηρεσιών ε, η, θεωρείται απειλή απέναντι σε κάποιους γείτονες. Δεν είναι μόνο η παγκοσμιοκίνδυση ο κίνδυνος και απειλή, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδατε ότι συζητήσαμε την οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων, ε, για την ελευθερή κυκλοφορία των εργαζομένων, ή ε, για την πιστοποίηση των προσόντων. Δεν τολμώ να πω ότι έχουμε αρκετή εμπειρία. Χρειάζεται μία τριετία να συλλέξουμε την εμπειρία και μετά να αξιολογήσουμε. Είναι πολύ νωρίς ακόμα για την καινοτομία. Πώς μετράμε την καινοτομία. Πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι υπάρχουν διάφορα είδη καινοτομία που είναι σημαντικά για την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Υπάρχει και πιο ριζική μορφή καινοτομία για τις ε, καινούργιες εταιρείε, αλλά υπάρχουν και πολλές καινοτομίε που είναι λιγότερο δραστικές, λιγότερο δυναμικές, αλλά εξίσου σημαντικές για το μέλλον της καινοτομία και της εφευρές. Όταν προσπαθούμε λοιπόν να μετρήσουμε και να αξιολογήσουμε την καινοτομία, θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα διάφορα είδη και πώς διασυνδέονται μεταξύ τους τις καινοτομίες. Γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε πανευρωπαϊκά πρότυπα, benchmarks ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακριβώς για τις πολύ νέες μορφές ε, καινοτομίας που είναι σπάνιες και αναδύονται ε, έτσι σποραδικά. τώρα, ποιες είναι οι ιδεώδεις πολιτικές, τι δουλεύει καλά και τι δεν δουλεύει, τι λειτουργεί καλά σας ετοιμάζουμε μια έκθεση, θα προσπαθήσω να, βάλω μερικά στοιχεία σχετικά εκεί. Γνωρίζουμε ορισμένα μόνο, όχι πάρα πολλά για τα όσα έγιναν, γιατί δεν γίνεται αρκετή αξιολόγηση στα μέσα και τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε. Πάντως κάποια στοιχειώδης έχει γίνει και μπορούμε να την αξιοποιήσουμε για το τι λειτουργεί καλά και τι λιγότερο καλά. Θα πρέπει να έχουμε πάντα τους σωστούς στόχους και τα προβλήματα να, εντοπίζουμε τα ε, προβλήματα που εμποδίζουν την πρόσβαση σε κονδύλια. Θέλετε να προσθέσετε τίποτα, κύριε Ανίδη. Ε, αναφορικά με τα ζητήματα της διοικητικής απλούστευσης, νομίζω ότι η πιο ε, ολοκληρωμένη, εξαιρετικά σημαντική μάλλον πρόταση είναι η ανάπτυξη one-stop shops για τον επιχειρηματία. Έχει αποδειχθεί από την ε, εμπειρία ότι στο μέτρο που μπορούν, ε, που μαζευτούν όλες οι διαφορετικές υπηρεσίες ή η γραφειοκρατία που θα πρέπει να παρακολουθήσει ο επιχειρηματίας για την οποιαδήποτε επιχειρηματική δουλειά που θέλει να κάνει σε ένα σημείο, ε, μπορεί να επισπεύσει πάρα πολύ τον απαραίτητο χρόνο. Τώρα, όσον αφορά τι ε, επενδύσει, είναι προφανέ ότι δεν, ισχύει, δεν ισχύουν τα ίδια πράγματα για όλε τι χώρε τη Ευρώπη. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι η γενική κατεύθυνση θα πρέπει να είναι μια προσπάθεια να ενισχυθούν ε, ε οι μικρομεσαίες επιχειρήσει, να γίνουν περισσότερο ένταση κεφαλαίου για τον λόγο ότι στην αντίθετη περίπτωση σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία θα υπάρχει μια μόνιμη πίεση στου μισθού, στην οποία δεν μπορεί η Ευρώπη να ανταγωνιστεί με χωρί χαμηλότερου κόστου. Τέλο, για τη χρηματοδότηση, θα λέγω ότι μπορούμε να εξετάσουμε και κάποια πράγματα που συνήθω τα αφήνουμε λίγο στην άκρη. Για παράδειγμα, 50% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα για να κάνουν ε, ε, επένδυση δεν προσφεύγουν στον τραπεζικό δανεισμό, αλλά προσπαθούν να τα βρουν από ίδια κεφάλαια. Άρα μέτρα πολιτική που να ενισχύουν αυτού του τύπου τη δυνατότητα δημιουργία ενό κεφαλαίου στο εσωτερικό τη επιχείρηση και στη συνέχεια να επενδυθεί, με φορολογικέ απαλλαγέ κλπ. θα ήταν αρκετά χρήσιμα. Äh, ευχαριστώ. Ε, συνάδελφοι Μπένσεν και Περβάνς. Όχι, πρώτα ο κύριος Μπένσεν, Μπένσεν και μετά η ε, Περβάνς. Under den første del af høringen i dag hørte vi om, hvilken øh, effekt af krisen... Er. Σας ευχαριστώ. Σήμερα ακούσαμε ποιο είναι ο αντίκτυπο τη κρίση στι μικρομεσαίε επιχειρήσει ε, και σε αυτή τη φάση το ερώτημα που μα απασχολεί είναι τι μπορούμε να κάνουμε. Θεωρώ πως είναι σαφές από τα όσα ακούσαμε σήμερα πως ε, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η χρηματοδότηση για τις ε, μικρομεσαίες μας επιχειρήσεις. Και είναι σαφές πως όντως χρειάζονται πόρους για να μπορέσουν να λύσουν τα προβλήματά τους. Τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε ως πολιτική του Ευρωκοινοβουλίου εμείς έχουμε μία οδηγία για τις πληρωμές, στην οποία ορίζονται ποιες είναι οι διατάξεις όταν δεν υπάρχουν πληρωμές, όταν δεν γίνονται οι πληρωμές. Η οδηγία αυτή είναι πολύ συγκεκριμένη όσον αφορά τους περιορισμούς στο business to business, θέτει κανόνες πολύ συγκεκριμένους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όταν έχουν να κάνουν συναλλαγές μεταξύ τους. Τώρα υπάρχει μια τάση των μεγάλων να καταπίνουν τις μικρές ή να τις αφήνουν στην άκρη, ε, πίσω. Ε, τι θα γίνει λοιπόν, αυτοί, αυτοί οι κανόνες δεν θα χρησιμοποιηθούν και για τις συναλλαγές business to business. Υπερβάω τώρα. important. Σας ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντικό, συμπεριλαμβανομένων των πρωτοβουλειών της ε, Ισπανικής Προεδρίας, που σκοπεύει να ανοίξει την ε, συζήτηση. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια συζήτηση που τώρα γίνεται στην Ισπανία. Θα δούμε αν θα φτάσει και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι ακριβώ ένα από του δρόμου που μπορεί να αναπτύξουμε. Να δούμε λοιπόν πώ ε, η μικρή ομεσαία επιχείρηση εκτίθεται απέναντι στην πτώχευση και στα ίδια περιουσιακά στοιχεία, σε, ε, ε, εκτίθεται δηλαδή σε μια κατάσταση ευάλωτη. Ίσως λοιπόν μια κοινή, ένας κοινός προβληματισμός από αυτού θα έπρεπε να γίνει. Και τώρα, να σας πω δύο παρατηρήσεις. Καταρχήν, όλοι συμφωνούμε ότι θέλουμε να έχουμε μικρομεσαίες που να μπορούν να αναλάβουν κίνδυνο και να δημιουργούν θέσεις απασχόλησης. Και έπειτα, ένα από τα πράγματα που πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν για το μέλλον είναι να βελτιωθεί και να, μείνει σε μια, και να παραμείνει σε σταθερό επίπεδο το επίπεδο κατάρτισης. Πολύ συχνά όταν το λέμε αυτό με εκπροσώπους των ε, ΜΜΕ μας λένε ναι, εσείς μας επιβάλλετε διάφορες υποχρεώσεις για κατάρτιση και πώς θα τα καταφέρουμε να έχουμε τρεις υπαλλήλους όλους και όλους κτλ. κτλ. Μήπως λοιπόν χρησιμεύει αυτή η ιδέα του κυρίου Κομφεράτη που είπε να μπουν να συνεργαστούν μεταξύ τους οι ΜΜΕ μπας και τα καταφέρουν. Ας είμαστε δημιουργικοί δηλαδή να έχουν μια διάρκεια ζωής πιο μόνιμη. Και έπειτα, έχουμε δει τις λεπτομέρειες για να καταλάβουμε τι πρέπει να διορθώσουμε. Γιατί θυμάμαι εκείνη τη συζήτηση που είχαμε όταν υιοθετήσαμε την Βασιλεία 2 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ένας από τους κανόνες που υιοθετήσαμε ήταν η ιδέα ότι η τράπεζα πρέπει να δικαιολογήσει δημόσια την άρνηση και τα κριτήρια με βάση τα οποία δίνει πιστώσεις. Εγώ ανέκαθεν πίστευα πως αυτό ενοχλούσε την, κατά, την, την ποιότητα τη συζήτηση που θα μπορούσε να έχει με τη ΜΜΕ μια τράπεζα. Πιστεύετε πως πρέπει αυτό να διορθωθεί όσον αφορά την πρόσβαση των μικρομεσαίων στην χρηματοδότηση. Σε αυτή τη συγκεκριμένη νομοθεσία Βασιλεία 2 υπάρχουν σημαντικά ζητήματα που θα πρέπει κατά την άποψή σα να επανεξετάσουμε. Κυρία Φόγγελερ, θέλετε να αρχίσετε εσεί Καλέ ερωτήσει, αλλά δύσκολε στην απάντησή του όλε. Ε, θα προσπαθήσω να απαντήσω ταυτόχρονα. Το σημαντικότερο που ήθελα να πω είναι ότι όλα τα εργαλεία, είτε είναι εκπαίδευση, είτε είναι δίκτυα, είτε είναι χρηματοδότηση, ε, θα πρέπει να τα δούμε διαφοροποιημένα στο εσωτερικό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, γιατί άλλες ανάγκες μπορεί να έχουν οι εταιρείε ε, ανάλογα με αυτά τα τρία. Ο συνάδελφός μου θα απαντήσει ε, για τις ανάγκες μιας μέσης, ας πούμε, μικρομεσαίας επιχείρησης, αλλά αυτές οι νέες καινοτόμες επιχειρήσεις, Young Innovative Companies, ε, είναι διαφορετικές και στα τρία αυτά στοιχεία. Ό,τι πολιτική, πάντως ανεξάρτητα αποφασίζεται, χρειάζεται τέτοια διαφοροποίηση. Ιδιαίτερα για τη χρηματοδότηση, ως παράδειγμα. Είναι πραγματικά διαφορετικές ε, οι ανάγκες, το κεφάλαιο κινδύνου, ε, τα τραπεζικά δάνεια. Είναι πολύ διαφορετική η κατάστασή τους. Και τι μπορεί να γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα μιλήσει περισσότερο για τα τραπεζικά δάνεια ο συνάδελφος, αλλά για τις νέες καινοτόμες επιχειρήσεις. Αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε μια αγορά διαχείρισης κεφαλαίου κινδύνου σταθερή και βιώσιμη, που να χρηματοδοτεί ακριβώς τέτοια σχέδια θα πρέπει να γίνει μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή είναι η κρίσιμη κλίμακα που χρειάζεται. Είναι πολύ μικρό το τοπικό επίπεδο για να εξασφαλιστεί μια τέτοια λειτουργία. Το σωστό επίπεδο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύω. Ευχαριστώ. Yes, of Για το θέμα των πληρωμών, ναι, θα ήταν απόλυτα απαραίτητο οι συναλλαγέ μεταξύ επιχειρήσεων να τυχάνουν τι ίδιε αντιμετωπίσει όπω οι συναλλαγέ μεταξύ επιχειρήσεων και κυβερνήσεω. Αλλά άμα δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη συζήτηση στο Συμβούλιο, βλέπουμε ότι οι μεγάλες πληρωμές ε, του δημοσίου τομέα ανεμπιστοποιούνται με τέτοιο τρόπο που δεν είμαι καθόλου αισιόδοξο ότι όλα αυτά θα είναι χρήσιμα για αυτά. Επίσης, κανένα από τα όργανα έχει ξεκινήσει με το πρόβλημα B2C, δηλαδή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, που προσφέρουν υπηρεσίες στους ιδιώτες, θα πρέπει να δούμε γιατί οι ιδιώτες δεν πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν έγκαιρα. Κατάρτιση Συμφωνώ ότι οι ΜΜΕ βρίσκονται σε πάρα πολύ συγκεκριμένη κατάσταση όσον αφορά την συνεχή ε, κατάρτιση. Γιατί είναι μικρές οι επιχειρήσεις. Δεν μπορούν να έχουν έναν που να είναι πλεονασματικός και να μπορούν να το στείλουν κάπου να εκπαιδευτεί. Εκτός αυτού υπάρχει ο κίνδυνος ότι ο αναγνωριστής θα τους τον πάρει, ίσως προσφέροντας κάτι παραπάνω. Και το καλύτερο λοιπόν είναι όταν πάνω από το επίπεδο της επιχείρησης, σε κάποια περιφέρεια, σε κάποιο τομέα, να υπάρχουν κοινά προγράμματα κατάρτισης για όλους τους τομείς ε, του ε, ΜΜΕ, οργανωμένοι από τους κοινωνικούς εταίρους, από τα εμπορικά επιμελητήρια, οποιοδήποτε. Αυτό είναι πολύ πιο αποτελεσματικό. Και μια τελική πρόταση για τη χρηματοδότηση. Αυτό που λέτε, που θέλετε να προτείνετε, είναι να υποχρεωθούν οι τράπεζες να δίνουν ε, δάνεια στις ΜΜΕ. Από την άλλη μεριά και οι τράπεζες πρέπει να έχουν την επιλογή να πάρουν απελάτη να μην το πάρουν. Αλλά εντάξει, είναι μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με χρηματοδότηση από δάνεια στη, σε όλες τις χώρες. Είναι ότι αυτή τη στιγμή τα φορολογικά συστήματα υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις κατά κάποιο τρόπο να χρηματοδοτηθούν από δάνεια. Θα πρέπει λοιπόν όταν συζητάμε τις ΜΜΕ να συζητήσουμε και τα εθνικά φορολογικά συστήματα, δεν θα φτάσουμε πουθενά. Ναι, ένα σύντομο σχόλιο γιατί με κάλυψαν οι προηγούμενοι για τα κυριότερα ζητήματα. Υπάρχει ένα πρόβλημα πολιτισμικό θα έλεγα σε πολλές περιπτώσεις τουλάχιστον στην Ελλάδα όσον αφορά τη δημιουργία δικτύων επιχειρήσεων. Οι επιχειρηματίες για κάποιο λόγο δεν θέλουν, ε, φοβούνται να συνεργαστούν μεταξύ τους. Προφανώς η απάντηση σε αυτό δεν μπορεί να είναι, δεν υπάρχει μία μόνο απάντηση. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι πάρα πολύ σημαντικό ρόλο μπορούν να παίξουν τα κέντρα προώθησης καινοτομία. Όταν δηλαδή μια μονο απαντηση σε καθε περιπτωση νομιζω οτι παρα πολυ σημαντικο ρολο μπορει να παιξουν τα κεντρα προθεση καινοτομια οταν δηλαδη μια επιχειρηση απευθυνεται σε μια ε, διοικητική μονάδα προκειμένου να τη βοηθήσει για να φτιάξει ένα business plan ή να μπορέσει να διαμορφώσει ένα, το μέλλον της το επόμενο, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή η μονάδα να μπορεί να έχει τη δυνατότητα και τη γνώση να τη διασυνδέσει με αντίστοιχε διαδικασίε, είτε κάθετα είτε οριζόντια, και να μπορέσει να αναπτύξει τα επιχειρήματα υπέρ αυτή τη ε, κατάσταση, ελπίζοντα ότι φυσικά ο επιχειρηματία, το οποίο είναι τελευταία απόφαση είναι δικιά του, θα ε, επιλέξει τέλο πάντων να μπει σε αυτή τη ε, διαδικασία. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλο του γύρου των ερωτήσεων. Άννα Γιάννη και η Κέθινα έχουν ερωτήσει να προβάλλουν. Παρακαλώ, είστε σύντομοι. Thank Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Εγώ επανέρχομαι στα όσα υπόθηκαν και στα όσα υπογραμμίστηκαν και από την κυρία Μπέρες σε σχέση με του τους διάφορους κανονισμούς και τη σημασία τους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πράγματι, Mm. Όταν ε, μία τράπεζα μειώνει τον προπολογισμό της, είναι σαφές ότι θα πρέπει να κάνει κάποια συγκεκριμένα βήματα. Και άρα Ποιο ε, σε αυτή τη φάση θα ασχοληθεί με τι μικρομεσαίες επιχειρήσει ε, σε αντίθεση με τι μεγάλε. Εσείς θεωρείτε πω αυτή η πρόταση που έχουμε επιτάπητο ε, και που ακολουθούν και παρακολουθούν οι διάφορε ομάδε συμφερόντων ότι θα είναι βοηθητικέ, θα μπορέσουν όντω να στηρίξουν τι μικρομεσαίες επιχειρήσει με αυτή την πρόταση που θέλουμε εμεί να κάνουμε που την εμπνευστήκαμε και με τον, από τον Ομπάμα από τη δουλειά που κάνει σε σχέση με τις τράπεζες ή κινδυνεύουμε να τις ε, ζημιώσουμε. Και μιλήσατε για ομίλους, ventures, για την δομή των μικρών μεσαίων επιχειρήσεων για τα ευρωομόλογα, δηλαδή με λίγα λόγια, τι μπορεί να κάνει η Ένωση στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος. Μπορεί να βοηθήσει και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πιστεύετε πως υπάρχουν προοπτικές από αυτή την άποψη. Σας ευχαριστώ. Πάντα βιαστική είμαι. Ε, σε σχέση με το δίκτυο στήριξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μήπως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να αναπτύξει μια πιο σφαιρική αντίληψη, εικόνα, δηλαδή να βρει κάποιες ε, ομάδες μικρομεσαίων όπου οι επιχειρηματίες να μπορούν να φτιάξουν οι ίδιοι μια ομάδα επιχειρήσεων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε ε, κλίμακες επιχειρήσεων ή συμβουλές που μπορούν να τους δώσουν. Πιστεύω όπως εδώ εστιάζουμε όλοι στις καινοτόμες εταιρείες καθώς αυτές θεωρούμε πως θα μας οδηγήσουν εκτός της ε, κρίσης και σίγουρα η στρατηγική του 2020 εστιάζει την προσοχή στην καινοτομία και στην έρευνα και ανάπτυξη. Ε, Βλέπω, το ίδιο κάνουν και η ΕΠΑ και η Κίνα και η Ινδία και όλοι οι άλλοι. Μήπως πρέπει να φτιάξουμε λοιπόν μια κάποιος πιο ε, τυπική βάση, κάποια πιο τυπική πλατφόρμα που θα βοηθήσει τις καινοτόμες αναπτυχθούν. Ευχαριστώ. Για σύντομη απάντηση, κύριε Ούρμαν. Όσον αφορά το θέμα το τις κεφαλαϊκές απαιτήσει. Κανένας δεν ξέρει ακριβώς, ακριβώς τι σημαίνει. Ε, καταρχήν δεν είμαστε κατά κάποιων ε, φραγμών, κάποιων ε, Ξέρουμε ότι ας πούμε, σε μια έκρηξη θα είναι λίγο πιο ακριβό, αλλά σε μια ύφεση θα είναι βοηθητικό να έχουμε τέτοιες, τέτοια όρια. Ε, αν θέλουμε πραγματικά κάνουμε να κάνουμε στις, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το θα πρέπει να κάνουμε τέτοιο τρόπο ώστε οι τράπεζες να μην μπορούν να δείχνουν τι έχουν και τι δεν έχουν. Τώρα, αν θέλουμε να έχουμε κάποια προϊόντα, γιατί σε κάποιες χώρες ας πούμε ρυθμίστηκαν ως υψηλού κινδύνου, δηλαδή προϊόντα επισήμως χαρακτηρισμένα ως τριπλό α και έχουμε κάποιο ρυθμιστικό κεφάλαιο. Αν το ρυθμίσουμε αυτό, αν το μειώσουμε αυτό, μπορεί να φτάσουμε σε σταθεροποίηση. Δεν έχει νόημα να αυξάνονται οι κεφαλαιοκές απαιτήσει για τα ε, δάνεια έρευνας και ανάπτυξης. Δεν υπήρχε ποτέ κανένα πρόβλημα στο παρελθόν. Αυτές είναι τρεις γραμμές με βάση το τι περιμένουμε εμείς από την κεφαλαϊκή αγορά. Η κυρία Φόγελας, τι πρέπει να κάνουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι είδους προγράμματα. Αυτό που θα ήθελα να δω στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μετάβαση από την έρευνα στην καινοτομία και στο να φέρουμε νέες ιδέες στην αγορά. Τα περισσότερα προγράμματα βασίζονται σε δίκτυα ε, μεγάλα, αλλά οι μικρομεσαίες και οι νέοι επιχειρηματίες δεν συμμετέχουν εκεί στα μεγάλα δίκτυα. Εξάλλου, ε, ούτε είναι και το πιο αποτελεσματικό εργαλείο ένα τέτοιο μεγάλο δίκτυο για μια καινοτόμα επιχείρηση και ιδέες. Χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερη εστίαση στην καινοτομία ακριβώς, που δεν σημαίνει πάντα δικτύωση. Ε, μπορεί να είναι και μεμονωμένα ε, σχέδια. Ε, ερώτηση γιατί θα πρέπει αυτό να γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. διότι ακριβώς είναι η οικονομία κλίμακας για την επιλογή για να στέλνουμε μηνύματα σε εκείνους που θα επιλέγονται στα προγράμματα αυτά για να μπορεί να υπάρξει ένας μοχλός έτσι, ε, και να το χρησιμοποιήσουν ε, και στην ε, ιδιωτική αγορά της τράπεζες όταν απευθύνονται ως ατού ότι τους χρηματοδοτεί. Τώρα για τις ομάδες των επιχειρήσεων, οι clusters, στην αρχική φάση σίγουρα υπάρχει πρόβλημα να συνενώνονται οι επιχειρήσεις, αλλά θα πρέπει να είναι πολύ καλά σχεδιασμένες οι πολιτικές για να ε, συμπαρασύρονται και οι ιδιωτικές δυνάμεις που θα χρηματοδοτήσουν και θα κάνουν ανταγωνιστική αυτή την προσπάθεια. Δηλαδή με ανοιχτό τρόπο να είναι, με σύγχρονο τρόπο να είναι ανοιχτά αυτά τα κλάστερ. Ευχαριστώ. Τέλος, θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση που δείχνει το εξή. Είναι λογοπαίγνιο, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να μεταφραστεί εύκολα. Αλλά χρειαζόμαστε και αλλαγή νοοτροπίας για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Ξέρουμε όλοι τη σημασία τους. Ακούμε πολλά λόγια, αλλά στα συγκεκριμένα όταν ερχόμαστε στα έργα δυσκολευόμαστε. Στη Γερμανία λέμε ε, όταν ε, κινδυνεύει μια μεγάλη επιχείρηση επεμβαίνει ε, ο Ομοσπονδιακός Αετός που είναι το σύμβολο της κυβέρνησης. Όταν κινδυνεύει μια μικρή επιχείρηση έρχεται ο γήπας της πτώχευσης που είναι άλλο αρπακτικό αυτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και τους τρεις σας για την παρουσίασή σας, την παρουσία σας και για τις απαντήσεις σας ραντεβού την άλλη εβδομάδα στο Στρασβούργο στις 9 το πρωί στις 11 το μηνό, Θα συζητήσουμε τα δύο πρώτα θεματικά έγγραφα. Σας ευχαριστώ πολύ.